Um, Καλό σας απόγευμα. Αρχίζουμε γιατί νομίζω ότι το θέμα 1 είναι θέμα ουσίας και γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη διότι κανείς δεν έχει έγγραφα εκτός από αυτά που ίσως έχετε τυπώσει εσείς οι ίδιοι αυτό ε, γίνεται διότι το print shop είναι ακόμα στο Λουξεμβούργο και όλα τα έγγραφα έρχονται με φορτηγά, με αυτοκινητοπομπή από το Λουξεμβούργο. Ε, ζητώ συγγνώμη διότι θα περιμένατε να τα έχετε μπροστά σας ή θα ελπίζατε να τα πάρετε από το πίσω μέρος της αίθουσας. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική συνεδρίαση θα ήθελα λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη μετά τις ε, τελευταίες αλλαγές. Δεν θα εξετάσουμε την έκθεση Λάγκεν για τα παράγωγα σήμερα. Θα το συζητήσουμε στο Στρασβούργο στις 8 Μαρτίου το θέμα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, έγκριση των πρακτικών Τη συνεδρίασης τη 9 η και τη 10 η Νοεμβρίου, τη 23 η και τη 7 η Δεκεμβρίου. Έτσι κερδίζουμε χαμένο χρόνο. Έχετε σχόλια. Όχι, θεωρώ λοιπόν να εγκρίνεται. Σα Σας είπα ότι θα γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο την Δευτέρα, την 8η 8 στις 7. Και το θέμα θα είναι η έκθεση Λάγκεν για την αγορά παραγόγων κάθεση. Λάβετε το λοιπόν υπόψη ότι τότε θα συζητηθούν τα παράγωγα. Τώρα θα στραφούμε στο θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης που είναι το κοινό σύστημα του φόρου τη προστιθέμενης αξίας και ιδιαίτερα ε, το θέμα του invoicing. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπήρξαν πολλές τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Και θα κοιτάξω τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία από τις ε, τροπολογίες. Δέκα ήταν επιπρόσθετες τροπολογίες. Οι τροπολογίες που υπέβαλα αφορούν τη δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ενός συστήματος cash allowing βάσει των πληρωμών που έχουν ε, γίνει και που έχουν παραλευθεί αντί επί της βάσεως των, ε, του ΦΠΑ. Και αυτό θα δώσει ε, θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να δώσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη δυνατότητα προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να διαλέξουν την πιο κατάλληλη μέθοδο. Και αυτό βάσει και με την της ε, για τις μικρές επιχειρήσεις. Έχουν γίνει δύο τροπολογίες για να μειωθεί η περίοδος για την φύλαξη των τιμολογίων. Προτείνεται τα έξι έτη να μειωθούν είτε σε τρία ή σε πέντε έτη. Δεν πιστεύω ότι αυτή η περίοδος αποτελεί ε, τήρηση των ε, τιμολογίων αποτελεί ιδιαίτερη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, πόσο μάλλον όταν θα περάσουμε και στο ηλεκτρονικό σύστημα. Και μία έκθεση του TWC δείχνει ότι η περίοδος αυτής φύλαξης των τιμολογίων κυμαίνεται στα κράτη-μέλη μεταξύ 5 και 7 ετών. Η Επιτροπή θέλει να εναρμονίσει αυτό το διάστημα και νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη λύση ο μέσος όρος των 6 ετών. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τις επιχειρήσεις να φυλάνε ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αυτά. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με όσους υπέβαλαν σχετικές τροπολογίες και είμαι πρόθυμος να συζητήσω και μια περαιτέρω διευκρίνηση του κειμένου προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μεταφέρουν τα ετοιμολόγια αυτά στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας της ε, Κομισιόν να εξισωθούν τα τιμολόγια τα ηλεκτρονικά με τα τιμολόγια σε χαρτιά. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τις επιχειρήσεις και θα καταπολεμήσει και θέματα απάτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης παρακολούθησε τις εξελίξεις τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη ε, εξισώσει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια με τα τιμολόγια σε χαρτί και η ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικών υπογραφών δεν έχει οδηγήσει όμως σε μείωση των ε, περιπτώσεων απάτες. Είναι περίπτεη από κάποια άποψη η απέτηση για ηλεκτρονικές υπογραφές και για ηλεκτρονικά τιμολόγια. Επίσης, αναμένεται ότι με τα νέα αυτά εργαλεία θα περιοριστούν οι περιπτώσεις απάτης. Συμφωνώ λοιπόν με τις τροπολογίες του κυρίου Φόξ σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα φυσκάλες και θα θέλαμε να διευκρινίσουμε περαιτέρω την, διατύπωση της τροπολογίας τους προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν κατά την κατάρτιση της έκθεσής μου και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες στις τελευταίες ημέρες και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να ψηφίσουμε επί ενός κειμένου το οποίο θα μας βρει όλους σύμφωνους. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Οι σκιώδεις δεν ξέρω αν θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Φόξ. Να πάρει το λόγο και οι υπόλοιποι να μου πούν αν θέλουν να μιλήσουν κι αυτοί. you, Um... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα με τον τρόπο που έχει συνταχθεί η έκθεση και δεχόμαστε τις τροπολογίες οι οποίες θα μειώσουν τον γραφειοκρατικό φόρτο στις επιχειρήσεις τα κράτη-μέλη θα επιβάλλουν τους κανόνες εκεί όπου είναι αναγκαίο και η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τον εισηγητή στις τροπολογίες 1, 2, 6, 8, 10 και 11 διότι έτσι μειώνεται η γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις. Θα υποστηρίξουμε τις 3, ε, 5 και 7 3, 5 και 7, διότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες εκεί που κρίνεται σκόπιμο. Την ε, τροπολογία 4, η τροπολογία 4 ε, διασαφηνίζει την νομοθεσία. Την 9 όμως δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε, αν και θα ε, συνεργαστούμε με τον κύριο Κάσερ για να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τεχνικής αρρωγής έτσι ώστε να βελτιωθούν τα διοικητικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Αλλά δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται επιπρόσθετη χρηματοδοτική αρρωγή. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα κράτη-μέλη. Και με χαρά υποστηρίζουμε τις ε, τροπολογίες Taylor και Σμιτ που μειώνουν το φόρτο στις, ε, που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Ωραία. Κανένας άλλος ε, δεν ε, ζήτησε το λόγο. Θέλετε να μιλήσετε εξ ονόμας του Σμίτ, έχετε το λόγο. Είμαι ο Ραμόν Τεμόζα από τους φιλελευθέρους. Ο συνάδελφος δεν έχει φτάσει γιατί είναι στην Κοπενχάγη και έχει προβλήματα να φτάσει στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να σχολιάσω και να πω ότι ε, θα ήθελα ο κύριος Σμιτ να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία. Πρέπει να μειώσουμε τον ε, γραφειοκρατικό φόρτο για τις ΜΜΕ και ε, υπάρχουν δύο σημεία που όλοι Σμιτ σας ανέφερε στις προγενέστερες συζητήσεις διαφωνεί με την τροπολογία 3 αυτή είναι μία από τις δύο τροπολογίες που ε, τον βρίσκουν αντίθετο. Όσον αφορά την τρία, ο Όλη Σμιτ πιστεύει ότι θα πρέπει να κρατήσουμε το αρχικό κείμενο της Επιτροπής διότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος ότι ορισμένα κράτη-μέλη θα επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες στις επιχειρήσεις τους. Άρα αυτό αντιτίθεται με τον αρχικό, αρχικό του στόχο και δεν θα βοηθούσε να μειώσουμε την, τον γραφειοκρατικό φόρτο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ο Όλι Σμιτ αντιτίθεται και στην 14 της κυρίας Γκέρντι Στόχος της επιχειρήσης της οδηγίας είναι να μειώσουμε το φόρτο της τιμολόγησης, αλλά η κυρία Κέρντι πιστεύει ότι θα πρέπει να έχουμε το προηγμένο σύστημα ε, ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Στην Σουηδία υπάρχει εμπειρία ηλεκτρονικής τιμολόγησης χωρίς να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα πέραν της ηλεκτρονικής υπογραφής. Άρα οι τροπολογίες του Όλιτ Σμιτ μειώνουν το γραφειοκρατικό φόρτο για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα της ΜΜΕ, έτσι ώστε τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα τιμολόγια επιχάρτου να βρίσκονται, να θεωρούνται ισόβαθμα. Επίσης, θα πρέπει να μετατρέψουμε τις, τα τιμολόγια πιχάρτου σε ηλεκτρονικά βαθμία και αυτό θα ήθελα να προσθεθεί στα, στην τροπολογία, στις τροπολογίες του έτσι ώστε να ενδυναμώσει, να ενισχύσει τις προθέσεις του και θα πρέπει να δούμε τις βέλτιστες δυνατές πρακτικές έτσι ώστε ο καθένας να έχει την ελευθερία να αποφασίσει ό,τι θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη το... Έχουμε... Έχουμε πρόβλημα διαρμηνίας. Δεν καλύπτεται η γλώσσα σας. Μπορείτε να μας τα πείτε αγγλικά ή σε κάποια άλλη γλώσσα. Ό,τι προτίθεστε. Ε, δεν ζητήθηκε η δική σας γλώσσα. Ίσως την επόμενη φορά να σταθώ πιο τυχερός. Ήθελα να συγχαρώ τον κύριο εργασία του και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε κοινέ προσπάθειες έτσι ώστε ο γραφειοκρατικός φόρτος για τις ΜΜΕ είναι χαμηλότερος. Υπάρχουν 19 εκατομμύρια ΜΜΕ στην Ευρώπη και έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης να τις βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις ε, υπηρεσίες τους και να μην τις φορτώνουμε με υπηρεσίες που μπορούν να καλυφθούν από κάποιον άλλο, δηλαδή από τις ε, φορολογικές αρχές. Εγώ σκιώδης προσπάθησα να είμαι επικοδομητικός. Οι δικές μου τροπολογίες κινούνται προς την κατεύθυνση του να μειωθεί ο γραφειοκρατικός και διοικητικός φόρτος και θα ήθελα να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μου, ιδιαίτερα την 18, η οποία αφορά τη μετάφραση ορισμένων τιμολογίων στην επίσημη τους γλώσσα. Θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελεί γραφειοκρατικό φόρτο για τις ΜΜΕ και αν υπάρχει ανάγκη μετάφρασης θα πρέπει να αναλαμβάνεται από τις φορολογικές αρχές και όχι από τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό ε, αυτή είναι και η πρόθεση των ε, άλλων τροπολογιών και ελπίζω να την εγκρίνουμε την οδηγία εν τέλει. Ζήτω συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, γιατί δεν υπάρχει διερμηνία στη γλώσσα σας. Θα ήθελε κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Η Επιτροπή. Θέλετε το λόγο. Okay, yes, Mr. Ο κύριος Ντίμερ. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε για όλες τις ε, τροπολογίες που εντάσσονται πλήρως στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το στόχο της για την οδηγία, υπό την ευρία έννοια τουλάχιστον. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω όλες τις τροπολογίες, αλλά νομίζω θα βοηθούσε να διευκρινίσω κάποια θέματα για τρεις-τέσσερις ε, τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα, η μορφή αποθήκευσης των τιμολογίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει διαγραφή τώρα στο 247,2 της οδηγίας για το ΦΠΑ, βάσει της οποίας μπορούν να περάσουν στο σύστημα ηλεκτρονικών τιμολογίων οι επιχειρήσεις, ακόμη και αν το πρωτότυπο είναι επί χάρτου. Ε, νομίζω λοιπόν ότι οι τροπολογίε καλύπτονται από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρόνο διατήρησης, το χρόνο αποθήκευση ε, ε, από συγκριτικές μελέτες που έκαναν ε, τα κράτη-μέλη και βάσει άλλων εξωτερικών μελετών φαίνεται ότι μία εξαετής περίοδος ε, αντιστοιχεί στο μέσο όρο που προβλέπουν ε, προς το παρόν ε, τα κράτη-μέλη και για λόγους ελέγχου από πλευράς των φορολογικών αρχών ενδείκνεται αυτή η περίοδος. Η συρρήκνωση της περίοδου σε τρία χρόνια, παραδείγματος χάρη, θα μας ανησυχούσε. Το θέμα της εξέβρασης ε, ισορροπίας ανάμεσα ε, στις απαιτήσεις των φορολογικών αρχών ε, για να μπορούν να διεξάγουν τους ελέγχους και το δυσανάλογα μεγάλο διοικητικό άχθος θα έλεγα ότι όπως η τροπολογία 18 ε, λέει δεν μπορούμε να κάνουμε αυτόματη μετάφραση. Θα γίνεται κατά περίπτωση και αν συντρέχει ανάγκη η μετάφραση. Τροπολογία 19 τώρα που σχολίασε και ο κύριος Φόξ. Το θέμα της ηλεκτρονικής διοίκησης αναβάθμισε την διακρατική συνεργασία και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνούμε μαζί σας. Δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε κάτι σχετικό μέσα στην οδηγία για το ΦΠΑ, γιατί έχουμε το πρόγραμμα Φισκάλης και ισχύουν εξάλλου και άλλες οδηγίες για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάζα, θα θέλατε να κλείσετε το θέμα. Θα μιλήσω στη γλώσσα με τα Μαλτέζικα γιατί μου αρέσει που έχω διερμηνία και θέλω να έχω διερμηνία και στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Είμαι πολύ ικανοποιημένο με τις παρατηρήσεις που έγιναν. Και έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να καταλήξουμε σε συμβιβασμού για τις τροπολογίες αυτές που έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι βασικός στόχος ε, της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και δικό μου βασικός στόχος είναι να παρουσιάζονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιγότερα προβλήματα αναφορικά με τη γραφειοκρατία και θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ελευθερία να υιοθετήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες προκειμένου τελικά να διαμορφώσουν συστήματα πιο αποδοτικά από τα σημερινά. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος από το έργο των συναδέλφων μου και των σκιωδών της Επιτροπής μας. Σας διαβεβαιώ ότι την επόμενη φορά, όταν περάσουμε σε ψηφοφορία, η έκθεση αυτή θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των μερών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 16 Μαρτίου, στη συνάντηση της ομάδας, της ε, Επιτροπής. Και την, στην Ολομέλεια, στην, την 1η του Απριλίου. Και τώρα να περάσουμε στην ετέχεια έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας για το 2008 και να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους όσους υπέβαλαν τροπολογίες. Ε, πρόκειται για γνωμοδότηση και δεν μπορούσα να επεκταθώ. Υπάρχουν αυστηρά όρια. Χαίρομαι πάντως ε, γιατί έχουμε 18 ε, τροπολογίες που μπορούν να ενταχθούν στο κείμενό μου. Θα θυμάστε σίγουρα ότι όταν πρωτοπαρουσίασα το θέμα στην Επιτροπή, τόνισα τα σημεία που κατά τη γνώμη μου ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για τις δραστηριότητες του 2008 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα το θέμα της διαχείρισης ε, της κρίσης ε, και τις ε, προσπάθειες που κάνει για να επικουρήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, σχετικά με τη στόχευση των δανείων, την απορρόφηση των κονδυλίων, την ορθή μη χρήση των πιστώσεων της τράπεζας κτλ. Ε, και προσπάθησα να επικεντρωθώ σε αυτά τα τρία σημεία όταν συνέταξα το τελικό κείμενο και παρά τους περιορισμούς σχετικά με το μήκος της ε, γνωμοδότησης και τελικά δεν μπόρεσα να ασχοληθώ με την εξωτερική διάσταση των δραστηριοτήτων της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της ΕΤΕ. Παρόλα αυτά κατάφερα να αναφερθώ ακροφυγώς στο θέμα και σας είπα ότι ενέταξα στο κείμενο και κάποιες τροπολογίες. Ο κύριος Χάμπλουντ ε, Φερρυπίν είχε υποβάλει μια τροπολογία για την ε, ε, εξωτερική διάσταση και νομίζω ότι μετά από τις συζητήσεις μας τελικά ε, βρεθεί και μια ικανοποιητική συμβαστική λύση. Τώρα, δυσκολεύτηκα ε, να, να δεχτώ κάποιες ε, τροπολογίες διότι δεν ήταν ακριβή ή ορθά τα μεγέθη. Ε, που ε, συμπεριλάμβαναν. Τώρα σε σχέση με το σχόλιο της κυρίας Ζουλή για τη διαφάνεια προσπάθησα να καταλήξουμε σε συμβασμό αλλά δεν τα κατάφερα δυστυχώς. Οι διαφάνειε δραστηριότητε τη ΕΤΕ είναι κέρια σημασία, ναι μεν, αλλά ε, παρά ήταν ισχυρή αυτή η διατύπωση, παρά ήταν σκληρή. Ο κύριος ε, Μπέργκμαν ε, των Σοσιαλιστών υπέβαλε μια τροπολογία που μπόρεσα να δεχτώ. Ο κύριος Σάιστσεκ, τροπολογία 14 επίσης. Και από τους σοσιαλιστές, από τον κύριο Μπέργκμαν, είδα ότι ε, απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στο περιεχόμενο της τροπολογίας 15, όπου εξέφρασε επικρίσεις σχετικά με κάποια δάνεια της ΕΤΕ που διοχετεύτηκαν στην Ασία και στις χώρες ΑΚΕ. Προσπάθησα να διερευνήσω αυτό το θέμα και είδα ότι το ποσοστό αυτών των δανείων ή μάλλον αυτά τα δάνεια δεν συνιστούν και μία τάση. Έγιναν το 2008 ε, και στη συνέχεια ε, δεν επαναλήφθηκαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για μια σταθερή τάση που να απηχείται στις δραστηριότητες της ΕΤΕ για μακρόχρονικό διάστημα ε, συνέβησαν μόνο το 2008 σε μία χρόνια και άρα δεν πρέπει να δούμε βιαστικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ επίσης τον σκιώδη Σιγητή και είμαι πεπισμένη ότι με αυτές τις τροπολογίες θα γίνει και καλύτερο το κείμενό μου. Πρόεδρος, ε, ε, είπα κάποιος από τους ε, θέλει μήπως το λόγο, Ούντο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώ ο κύριος Μπέρμαν δεν θα μπορέσει να συμμετάχει σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Γι' αυτό λοιπόν τον αντικαθιστώ και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Συμφωνούμε ε, γενικά με, την ε, ευρύτερη, με τον ευρύτερο συμβιβασμό που κατάφερε να βρει σε ό,τι αφορά τους τομείς ε, στους οποίους θα πρέπει εκ νέου να την εντολή ε, εν ώψη και της νέας νομικής κατάστασης. Συμφωνούμε με τα δύο σημεία τα οποία έθιξε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δηλαδή θα πρέπει ε, αναλογικά και με τον κατάλληλο τρόπο να εκπροσωπείται στις γειτονικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστός καταμερισμός εργασιών σε ό,τι αφορά και την Τράπεζα Ανάπτυξης. Αυτά τα σημεία αποτελούν σημείο των ε, συμβιβασμών. Και δύο πτυχές αναφέρει η συγκήτρια σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες μας, ότι Κοιτάμε, όπως και στο παρελθόν, φυσικά την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι εκ παραλίλου θα πρέπει να ελέγξουμε και τις, ε, να μην παραμελήσουμε και τις ε, διεθνείς μας υποχρεώσεις και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξη της συζητήτρια σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες αυτές, σε ό,τι αφορά τώρα τις άλλες τροπολογίες σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις τροπολογίες των πράσινων. Καταλαβαίνουμε σε ό,τι αφορά την πιο σαφή πράσινη, αν θέλετε, κατεύθυνση που θα πρέπει να λάβουν οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το ελέγχουμε αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει και θα πρέπει να δούμε ποια επιτροπή θα είναι αρμόδια. θα πρέπει να διαμοιραστούν αυτέ οι αρμοδιότητε μεταξύ επιτροπή Οικονομικών και περιβάλλοντο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν επικοδομητικά να εργαστούμε επί τη έκθεση αυτή μέχρι τέλου. Äh, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας. Δεν είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που οι τροπολογίες μας ε, δεν υιοθετήθηκαν κατ' ουσία παρά το γεγονός ότι στην διαδικασία συμβιβασμών κάναμε κι εμείς κάποια βήματα προς τα εμπρός. Διαπιστώνω ότι κάποιες από τις τροπολογίες μας ιδιαίτερα είναι αυτονόητες στο πλαίσιο μιας κοινωνικής ε, οικονομίας της αγοράς, σε ό,τι αφορά δηλαδή και τη διαφάνεια, σε ό,τι αφορά ενέργειες με δημοσίους πόρους. Common sense, κοινή λογική είναι αυτές οι τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε δυσαρεστημένοι για το ότι δεν υιοθετήθηκαν τα σημεία αυτά. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει καταμερισμός εργασιών. Η Επιτροπή Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι αρμόδιες για τα θέματα αυτά και εκεί θα πρέπει να μείνουν τα θέματα αυτά, να μην τα πειράξουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ακολουθήσει η συζήτηση. Ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και νέες συζητήσεις, γιατί κάτι τέτοιο πραγματικά δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Μη πρόεδρος, κανείς άλλος, κάποιος άλλος από τους κοιόδης. Ο κύριος ε, Ντουκρέν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι παρόν. Θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Εντάχει, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική αυτή εργασία και ιδιαίτερα για την αγαστή συνεργασία που είχαμε για παροχή πληροφοριών και συζήτηση. Τώρα έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία για το τέλος του 2009. Θα ανακοινώσει ο πρόεδρος Μέιστα τα στοιχεία το τέλος της εβδομάδας μπορώ να σας δώσω δύο αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με την ανταπόκριση στην κρίση. Η τράπεζα προχώρησε στα 80 δις, 80 δις δανειοδότηση, που είναι υψηλότερο στοιχείο από το αναμενόμενο. Σε σχέση με τις ΜΜΕ, το ίδιο μπορεί να υποθεί και ίσως είναι και καλύτερα τα πράγματα, διότι η δανειοδότηση προς ΜΜΕ έφτασε στα 15 εκατομμύρια το 2009, που είναι το επίπεδο του 2007 επί 3. Ε, και ιδιαίτερα στα νέα κράτη-μέλη, στα οποία προσδίδουμε μεγαλύτερη σημασία, το στοιχείο αυτό πολλαπλασιάζεται επί 6 από το 2007. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε σχέση με τα ποιοτικά στοιχεία αυτής της δανειοδότησης, διότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε προσδώσει μεγάλη σημασία στο θέμα της διαφάνειας των συναλλαγών και της προσθέμενης αξίας. Υπάρχει η σύσταση να προωθήσουμε τα στοιχεία, αναδεκαδικό στοιχείο σε σχέση με τον δικαιούχο ή προς τις ΜΜΕ. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την κατάσταση της αγοράς, διότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στην τράπεζα που μεσολαβεί να αναλάβει το κίνδυνο. Ελπίζουμε λοιπόν να ε, αναλάβουμε περισσότερους κινδύνους και προωθούμε αυτούς τους μηχανισμούς για να μην φτάσουμε στην δανειοδότηση μέτζανιν, του ημιορόφου δηλαδή, ε, Επίση, υπάρχουν δύο άλλες συστάσεις να έχουμε ε, ένα ε, στοιχείο αποτίμησης σε σχέση με το, uh, σε σχέση με το επίπεδο μόχλευσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν θα ήθελα να κάνω πολλά σχόλια στις ε, τροπολίσεις στις τροπολογίες που πρότεινε η συνεργαζόμενη μας Επίτροπη, διότι υπάρχουν ορισμένες πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές που δεν μπορούμε να αναλάβουμε εμείς, αλλά εσείς. Θέλετε να επανέλθετε. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους από την ομάδα Πρασίνων και Σοσιαλιστών που συμμετείχαν στην ε, σημερινή μας συζήτηση. Δεν διαφωνούμε. Οπωσδήποτε θα πρέπει να αναφερθούμε στην κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Είναι όντως σημαντικό. Πιστεύω δε ότι αντέδρασε καλά και λογικά η Ευρωπαϊκή Τραπεζά Επενδύσεων στην κρίση. Το πρόβλημα ε, έγκυτο στην ε, διατύπωση των κάποιων τροπολογιών Δηλαδή μπορεί να δώσουμε την εντύπωση ότι οι περιβαλλοντικές ε, και οι κοινωνικές ε, πτυχές δεν ελήφθησαν δεόντως υπόψη από την τράπεζα. Αυτό δεν ισχύει. Η διαφάνεια έχει κέρια σημασία και, και θεωρώ ότι η ε, εκταμίευση ε, ενωσιακών ε, κονδυλίων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Είτε μιλάμε για την ΕΤΕ, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο φορέα. Ε, προς το παρόν ε, είναι αδιαφανής η διαδικασία, λένε κάποιες τροπολογίες. Γι' αυτό έχω πρόβλημα με την διατύπωση. Ε, σας υπέβαλα μια συμβαστική πρόταση, δεν μπορέσατε να την εγκρίνετε. Τέλος πάντων νομίζω ότι ξεκινήσαμε σε να ακολουθούμε τη σωστή οδο παρόλα αυτά. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου. Ε, και μετά στις 15 Μαρτίου στην Επιτροπή μετά θα περάσει από την Ολομέλεια. Εκτός και αν γίνει κάτι αναπάντεχο. Περνούμε τώρα στο σημείο 7 μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσιοοικονομικών για μια ε, οικονομία σε ανάκαμψη. Λίαν Πανκόκ, θα μας παρουσιάσετε την ε, πρότασή σας. Merci, Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή μας επιτρέπει να επανέλθουμε σε δύο από τα βασικά διδάγματα της κρίσης ως προς την επίπτωση που είχε επί των δημοσιοοικονομικών. Το πρώτο δίδαγμα έχει σχέση με τον κόντρα αντικυκλικό ρόλο που είδαμε στην κρίση τις δράσεις των κρατών και που εστέφθη με επιτυχία, αν μπορούμε να το πούμε. Ε, βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί τα δημοσιοοικονομικά είναι ακόμη σε επισφαλή κατάσταση. Δεύτερον, οι αγορές και οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης αντιμετωπίσαν ιδιαίτερες δυσκολίες ε, λόγω του ότι εκτροχιάστηκαν πολλά παράγωγα τον περασμένο χρόνο και δυσκολεύτηκαν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο που ενέχει η κατοχή των κρατικών ομολόγων. Πάει το μυαλό μας στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι το ελληνικό πρόβλημα έχει μεγάλη σχέση με την ίσπραξη ε, των φόρων. Αλλά δεν μας έρχεται στο μυαλό η Ισπανία που είναι ένας από τους καλύτερους μαθητές ε, σε σχέση με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ε, που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ισπανία προφανώς υφίσταται υπεραξιολόγηση κινδύνου που συνδέεται με την κατοχή κρατικών ομολόγων από πλευρά των αγορών. Οπότε, με αυτή την έκθεση μπορούμε λίγο να αποστασιοποιηθούμε για αυτά τα δύο βασικά ζητήματα για να βελτιώσουμε την ε, ε, διαχείριση του προπολογισμού στο μέλλον και ίσως και να επικουρήσουμε αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ούτως ώστε να κάνουν πιο αποτελεσματικά τις αξιολογήσεις ε, των δημοσιοοικονομικών. Για την δημοσιονομική πολιτική προτείνει η έκθεση να ε, μείνουμε μέσα στο πνεύμα της ε, αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας ε, που χρονολογείται το 2005 που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αποκλίνουν από τα κριτήρια του Μαστρίχτ όταν ισχύουν έκτακτες συνθήκες και κυρίως όταν υπάρχει ύφεση. Αυτό εξάλλου επέτρεψε στην Επιτροπή να διαχειριστεί την κρίση. Η αναθεώρηση του συμφώνου είναι ένα δείγμα ε, ρεαλισμού. Αν αποστασιοποιηθούμε και δούμε θεωρητικά το ζήτημα, βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια που προτείνονται μέσα στην έκθεσή μου ούτως ώστε ε, η αντικυκλική μεταχείριση των δημοσιονομικών ελλημάτων να είναι αποτελεσματική. Και είδατε με την κρίση, το αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτή είναι η ορθοί δημοσιονομικοί κανόνες. Τι μπορούμε να προτείνουμε λοιπόν. Παραδείγματο χάρη, όσο οι παραγωγικέ ικανότητε ε, υστερούν σε σχέση με την κανονική ψαλίδα του, ψαλίδα που βάσει του μακροοικονομολόγου κυμαίνονται από το 75 έω το 85% των ικανοτήτων. Αν λοιπόν τοποθετούνται ε, κάτω από αυτήν την ψαλίδα, θα μπορούσαμε να προτείνουμε την διατήρηση των μέτρων στήριξης και τη διατήρηση των μη συμβατικών μέτρων, έτσι θα αποκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν όταν φτάσει στην κανονική ψαλίδα χρήσης των παραγωγικών ικανοτήτων της οικονομίας, δηλαδή στο 80-85%, ε, τότε μπορούμε να ε, προτείνουμε το εξή. Τα πλεονάσματα του πρωτογενούς προϋπολογισμού που θα έχουν προκύψει να τα χρησιμοποιήσουμε για την αποπληρωμή του χρέους και άρα να βρούμε δημοσιονομική, να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό ε, και βέβαια με την προοπτική της πλήρους απασχόλησης ταυτόχρονα. Αυτοί οι κανόνες είναι πολύ συγκεκριμένοι και χάρη σε αυτούς δυνάμεθα να κάνουμε και συστάσεις για τη στρατηγική εξόδου, exit ε, strategy. Ξέρετε ότι συζητείτε το θέμα. Εάν το 2010 ε, Αναστείλουμε τα μέτρα στήριξης και επανέλθουμε σε πολιτικές εξόδου. Ε, καταλαβαίνουμε τι, ότι σήμερα στην Ένωση των 27 έχουμε χαμηλότατες παραγωγικές ικανότητες, 70%. Πολύ κάτω από την, ε, ε, από την κανονική ψαλίδα. Οπότε αν αναστείλουμε όλα τα επανομαζόμενα μη συμβατικά μέτρα, γρήγορα θα βυθιστούν και πάλι οι οικονομίες μας ε, στην ύφεση. Εν τη αυτή περιπτώση να προτείνουμε τη διατήρηση των μέτρων στήριξη όσο υπάρχει ε, χαμηλή χρήση των παραγωγικών ικανοτήτων για να ε, βρούμε μια διέξοδο από την κρίση μέχρι να φτάσουμε στην κανονική χρήση των παραγωγικών ικανοτήτων. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου, ένα σημαντικό στοιχείο της έκθεσης. Επίσης, πώς θα αποσβεθούν οι κραδασμοί στην κοινωνία για τις δημόσιες δαπάνες, αλλά όχι μόνο. Μέσα στις δημόσιες δαπάνες υπάρχουν οι, κρατικές, οι κοινωνικές δαπάνες. Και αντίθετα με τη ΣΥΠΑ, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο κατάφερε να αποσβέσει τους κραδασμούς με εξαιρετικό τρόπο μετά την κρίση. Και χάρη σε αυτό το πρότυπο οι οικονομίες μας ανέκαμψαν σχετικά γρήγορα. Και σας παραπέμπω και στη συζήτηση που θα κάνουμε με τους ε, συναδέλφους μας από την Επιτροπή Κοινωνικών ε, Υποθέσεων ε, που καλούνται να συζητήσουν το θέμα του μέλλοντος που επιφυλάσσουμε στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Αλλά καλό θα ήταν να επιλεγεί η σωστή λύση για να προστατεύσουμε τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Δεύτερο θέμα της εκθεσής μου που επίσης μας απασχολεί όλους εδώ, το θέμα της βιωσιμότητας, μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημοσιοοικονομικών. Λοιπόν, ε, φυσικά πρέπει να προσδιορίσουμε ένα κριτήριο που να είναι συμβατό με αυτό το αντικυκλικό στοιχείο διαχείρισης των ελλημάτων του προϋπολογισμού που μόλις περιέγραψα. Μία προκατακτική παρατήρηση τώρα για να επισημάνω ότι δεν προβλέπεται στην οικονομία αδιαμφισβήτητο κριτήριο για να μετρήσουμε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οικονομικών. Οι οικονομολόγοι δεν ξέρουν να περιγράψουν τι, ε, τι σημαίνουν αυτά τα σταθερά ε, δημοσιοοικονομικά μακροπρόθεσμα. Ε, θα πρέπει να είναι το επιτόκιο δανειοδότησης ε, υψηλότερο από το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται το κράτος που προσφέρει για τα κρατικά ομόλογα. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Οπότε δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προτείνει ένα δίκτυο. Εμείς στην έκθεση προτείνουμε ένα δίκτυο μέτρησης της μακροπρόθεσμης ε, βιωσιμότητας δημοσιοοικονομικών δίκτυο συμβατό με την αντικυκλική αυτή η χρειά της διαχείρισης του προϋπολογισμού, πάντοτε μακροπρόθεσμα. Ο δείκτης λοιπόν αυτός θα έλεγα ότι είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα και στόχος του είναι να συμπληρώσει τους λοιπούς δείκτες της συνθήκης του Μάστριχ και του Συμφώνου Σταθερότητας εφόσον ε, υπάρχουν μέσα στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες, δύο είναι και θέλουμε το κριτήριο του ελλείμματο του προπολογισμού, το 3%, το περίφημο, έτσι θέλουμε να το συμπληρώσουμε με τον δείκτη του διαρθρωτικού ελλείμματο. Δηλαδή αφού έχουν εξουδετερωθεί οι επιπτώσει της οικονομική συγκυρία επί του ελλείμματο. Και το δεύτερο κριτήριο που προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, είναι το πόσο στο ε, διαρθρωτικού χρέου λόγος του κρατικού χρέου επί των στοιχείων του ενεργητικού που κατέχουν τα κράτη. Με αυτούς τους δύο δείκτε έχετε αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία, ούτω ώστε να μπορέσετε να εκτιμήσετε σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης, ε, ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια και οι οργανισμοί αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα και οι αγορέ και το ελεγκτικό συνέδριο που ε, θα κληθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση του δημοσίου χρέου όπω ζήτησε και η Περβάν Μπερέσε στην προηγούμενη εκθεσή τη δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσκομα. Έτσι, εμείς μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την ποιότητα του δημοσίου χρέους κυρίως με τη διεξαγωγή μελετών αντικτύπου και αξιολόγηση σε διαφόρων μέτρων που ανελήφθησαν, μέτρων στήριξης. Είναι απαραίτητο να γίνουν μελέτες αντικτύπου, διότι εάν Παρότι μάλλον στα περισσότερα κράτη-μέλη ελέγχουμε τα δημόσια οικονομικά, υπάρχουν δαπάνες που έγιναν ε, αυτή την τελευταία περίοδο για να τονωθούν οι οικονομίες, οπότε είναι απαραίτητο πέρα από τις δαπάνες των μέτρων στήριξης να γίνει αξιολόγηση όλων των δαπανών, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε χρηστά τα περί τα δημόσια οικονομικά μας. Και αυτό θα γίνει μέσα από τις μελέτες αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank um, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε το Ο κύριος Χόκμαρκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μας δίνει, ε, αφήνει χώρο μάλλον για συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να δηλώσω το εξή που είναι σημαντικό από τη δική μας ε, άποψη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή κατά της απασχόλησης, της ευημερίας και της ανάπτυξης ε, παρά τα ε, δημόσια οικονομικά τα οποία υποβαθμίζονται. Και αυτό αφορά και το δημόσιο έλλειμμα. Θα ήθελα να επιθυμίσω στην Επιτροπή ότι πέρσι είχαμε να κάνουμε με μία έκθεση σε σχέση με την πολιτική ανάκαμψης, όπου μπορούσαμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο τάσεων. Η σοσιαλιστική ομάδα ζήτησε μεγαλύτερες δαπάνες ε, πιο χαλαρούς κανόνες σε σχέση με το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή να υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια ε, δημόσιου ελλείμματος και σε σχέση με τη δημόσια χρηματοδότηση, αλλά οι σοσιαλιστές έχασαν. Διότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των δημοσίων οικονομικών και αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω προς ε, τον εισηγητή, δηλαδή πώς η σοσιαλιστική ομάδα και οι σοσιαλιστές ε, στην Ευρώπη ζήτησαν να υπάρχει ο ίδιος ρυθμός δαπάνης όπως τις είπα στην Ευρώπη, στην ε, Ισπανία, παντού. Τώρα όμως έχουμε τα αποτελέσματα. Στην Ισπανία έχουμε μεγάλο δημόσιο έλλειμμα και η ψηλή ανεργία που ανέρχεται σε ένα 20%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ε, διπλασιαστεί το δημόσιο χρέος και αυξανόμενο κόστος κάλυψης των επιτοκίων του δημόσιου χρέους. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κόστος, μια πολύ μεγάλη δαπάνη που αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Επειδή έχουμε υψηλότερα επιτόκια, και επειδή ο δημόσιος δανεισμός υποσκάπτει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αν δούμε τις δύο εναλλακτικέ των σοσιαλιστών, όπως εφαρμόστηκε σε ορισμένα κράτη-μέλη και τον πιο ε, περισταλτικό τρόπο, βλέπουμε τα αποτελέσματα και είναι εύκολο να κρίνει κανείς τι είναι καλύτερο χαμηλότερη ε, δημόσια χρηματοδότηση, χαμηλότερα επιτόχια, χαμηλότερη χρηματοδότηση γενικά και πολύ υψηλή ανεργία. Αυτά είναι τα στιγνά στοιχεία, διότι και οι δύο εναλλακτικές εφαρμόστηκαν έμπρακτα και είναι εύκολο να κρίνει κανείς. Γι' αυτό έχει σημασία τη στιγμή που προχωράμε με μία συζήτηση για μία στρατηγική εξόδου, θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη του να προχωρήσουμε να μειώσουμε το έλλειμμα στα διάφορα κράτη-μέλη πρωτίστως, πρωταρχικά. Γιατί διαφορετικά θα είμαστε στην ίδια κατάσταση, οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Ευρώπη τη δεκαετία του 70. Χρειαζόμαστε έλεγχο, πρέπει να έχουμε συνολικό έλεγχο των δημοσίων δαπανών, διαφορετικά υποσκάπτουμε το οικονομικό μας μέλλον θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όταν μειώσουμε τα δημόσια ελλείμματα, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, θα πρέπει να ανακάμψει η οικονομία α, αναπτύσσοντας τις προμήθειες, να αυξήσουμε τις δυνατότητες για επενδύσεις και για συναλλαγές ε, διασυνοριακής φύσης και για νέες αγορές οι οποίες θα πρέπει να ανακύψουν. Σε σχέση τώρα με την βιωσιμότητα, τη μακροχρόνια βιωσιμότητα. Νομίζω είναι πολύ εύκολο να δούμε ότι τα ελλείμματα που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη-μέλη, και δεν αναφέρομαι στα πιο δύσκολα παραδείγματα, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αύξησης δημοσίων δαπανών όταν δεν ελέγχουμε τα δημόσια οικονομικά. Δηλαδή αυτό που μας πλήττει σήμερα είναι τα δημόσια λύματα ορισμένων κρατών μελών. Αυτό πλήττει το ευρώ και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Γιατί ισχύει αυτό. Διότι πολλά κράτη-μέλη είχαν πολύ υψηλά ελλείμματα πριν επέλθει η οικονομική κρίση. Και νομίζω ότι όταν κοιτάμε προς τα εμπρός θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα ορίσουμε νέους κανόνες του παιχνιδιού έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα μακροχρόνια στις ε, μακροχρόνιες ε, ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους χειρότερους, τους πλέον δυσίωνους καιρούς. Ένα από τα λάθη μας είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη, τα περισσότερα, αυτό ακριβώς έκαναν, δεν προέβλεψαν τους δυσίωνους καιρούς με τα υπέρογκα δημόσια ελλείμματα. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να δημιουργούμε αυταπάτες σε σχέση με την αξιολόγηση του δημοσίου ελλείμματος, διότι μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο αξιολόγησης ε, του δημοσίου ελλείμματος στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Το ζήτημα όμως είναι τι επιτόκια θα πρέπει να καταβάλουν οι πολίτες όταν οι κυβερνήσεις δεν έχουν πια τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών, των δημόσιων δαπανών. Αυτό το βλέπουμε σήμερα σε πολλά κράτη-μέλη και μπορώ να ε, πω στον εισηγητή ότι δεν είμαστε καθόλου ευτυχείς. Είναι δική μας ευθύνη να ορίσουμε τα θεμέλια για, μια, για υγιή δημόσια οικονομικά, για ε, δυνατότητες, για νέα απασχόληση, για πρόθεση των οικοκυριών και για ανάπτυξη των οικοκυριών και αυτές τις τροπολογίες θα προωθήσουμε. Θα δούμε πρώτα με τους σκιώδεις πριν ε, μιλήσουν τα άλλα μέλη. Hegland, Καλ Hegland. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ καταρχάς ε, την προσέγγιση σου σε ό,τι αφορά την ε, στρατηγική εξόδου, σε ό,τι αφορά την έξοδο δηλαδή από την ε, δύσκολη αυτή κρίση. Και επίσης θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Χακμάρκ. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και εν ώψη των τελευταίων εβδομάδων και των εξελίξεων των τελευταίων εβδομάδων. Καλά θα ήταν λοιπόν να αποτυπωθούν όλα αυτά στην τρέχουσα έκθεση. Ο εισηγητής αναφέρθηκε στην προσέγγιση των δημοσιονομικών που θα πρέπει να ακολουθηθεί και αυτό είναι πολύ ωφέλιμο σε συνδυασμό δε με το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες θα πρέπει να υπάρξει περιορισμός των εξόδων, των δαπανών. Κάπως θα πρέπει να εξέλθουμε από την κρίση αυτή. Και γι' αυτό θεωρώ ότι σωστό θα ήταν να γίνουν κάποιες ε, προσαρμογές στην έκθεση. Ασφαλώς, ανακύπτουν πολιτικά ζητήματα. Είναι μάλιστα και φιλοσοφικό το θέμα του κατά πόσο και πώς θα εξέλθουμε τις κρίσεις. Κοιτώντα μάλιστα και τα αριθμητικά στοιχεία για κάποια κρατημέλη σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι θα προκύψει μακροπρόθεσμα ενδεχομένως έλλειμμα. Και θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι ποσοστό θα απορροφηθεί. Στα μισά κράτη-μέλη, ωστόσο, έχουμε φτάσει στο maximum. και θα ακολουθήσουν και τροπολογίες από την ομάδα μου. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ανέφερε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ασφαλώς σε πάση θυσία το κράτος πρόνοιας. Φυσικά μπορούν να γίνουν περικοπές στα δημοσιονομικά στους ε, δημόσιους προπολογισμούς. Η κατάσταση ωστόσο είναι σοβαρή. Όπως σας είπα, σίγουρα αυτή η συζήτηση θα είναι ενδιαφέρουσα και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία, ο κύριος Κίκολτ. Ευχαριστώ για την έκθεση. Όντως. Θα έπρεπε να συζητήσουμε εις βάθος ε, τις λεπτομέρειες που αφορούν ε, τα δημοσιονομικά, την Ευρωζώνη. Υπάρχουν διάφορες επικαλύψεις, αν θέλετε, διάφορα κοινά στοιχεία μεταξύ των εκθέσεων αυτών. Ωστόσο, παραμένουν διαφορετικές ως εκθέσεις και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει διαφορετική συζήτηση. Καταρχάς, θα πρέπει σας ευχαριστήσω που προσπαθούμε να βάλουμε κάποια κάποιον ορθολογισμό δηλαδή στη συζήτηση, για να μην πούμε δηλαδή ότι το δημόσιο χρέο είναι καλό ή κακό, ότι οι δημόσιε δαπάνε είναι πολύ υψηλέ, πολύ χαμηλέ και ούτω καθεξή. Όχι δηλαδή να παρηχαρακώσουμε ιδεολογικά το θέμα, αλλά να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα κριτήρια. Και αυτό που μου αρέσει στην έκθεση και θα ήθελα να αποτυπώνεται και στη συζήτηση είναι να κοιτάξουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα, συγκεκριμένα κριτήρια. Αντί να επαναλαμβάνουμε διαρκώ ότι, για παράδειγμα, δεν πρέπει να είναι πολύ ψηλό το δημόσιο του χρέους. Για τον τρόπο τώρα που προτείνεται ως λύση πρέπει να σας πω ότι έχουμε αμφιβολίες ως πράσινοι. Τι πρόταση λοιπόν γίνεται. Η πρόταση που γίνεται είναι να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες μέχρι να φτάσει στο 85% το δυναμικό παραγωγής. Δηλαδή ο εισηγητής θέλει στον τομέα της ε, βιομηχανικής παραγωγής τα προϊόντα αυτά τα οποία καταστρέφουν τον πλανήτη να τονωθούν. Εμείς ως πράσινοι αυτό ακριβώς θέλουμε να μην γίνει όταν μιλάμε για το Green New Deal. να μην ε, φτάσουμε πάλι στο maximum την λάθος παραγωγής, των λάθος προϊόντων. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση. Γιατί τα θέματα της αναδιάρθρωσης της βιομηχανικής μας παραγωγής δεν τίθενται επαρκώς. Δεν κοιτάμε πώς παράγουμε προκειμένου να μην προκύψουν τελικά οικολογικά χρέη. Αυτή λοιπόν ότι η βασική αρχή ότι το δημόσιο χρέος μπορεί να έχει διάφορες πτυχές αυτή η αρχή δεν αποτυπώνεται στην έκθεση αυτή και γι' αυτό δεν ε, δυσκολευόμαστε να την αποδεχτούμε. Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε ποιο είναι το σωστό επίπεδο χρέους. Ποιο είναι το βιώσιμο επίπεδο χρέου. Αυτό δεν σε αμφισβήτηση. Αλλά αυτή η νομιμοποίηση τη δημόσιας δράσης είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα. όπου διακυβεύεται και όπου τίθεται σε αμφισβήτηση το δημόσιο χρέος οι πολίτε στη Γερμανία δεν αναφέρουν ότι το βασικό πρόβλημα είναι η οικολογική κρίση, η ανεργία, αλλά το επίπεδο του δημόσιου χρέους και το ενδεχόμενο να καταστεί ανίκανο προς δράση το κράτος. Θα πρέπει να λάβουμε λίγο πιο πολύ στα σοβαρά αυτή την ανησυχία και να μην απαντάμε μόνο με μακροοικονομικούς όρους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που σε ένα σημείο αναφέρεται στην οικολογική μεταρρύθμιση. Αναφέρει ωστόσο εκεί ότι οι απαραίτητες επενδύσεις θα πρέπει να προέλθουν από το δημόσιο κλάδο κυρίως. Ωστόσο εμείς θεωρούμε ότι το δημόσιο σκέλος θα πρέπει να ε, προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να υπάρχουν ιδιωτικές επενδύσεις στον ε, τομέα αυτό των οικολογικών μεταρρυθμίσεων. Άρα, στην αναδιάρθρωση της οικονομίας, στη μεταρρύθμιση της οικονομίας, δεν μιλάμε κατά κύριο λόγο για δημόσιες επενδύσεις. Όχι, θέλουμε απλά ένα σωστό πλαίσιο προκειμένου να προκύψουν μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και νομίζω ότι στο θέμα αυτό, στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επί μια λίγο διαφορετική ε, διατύπωση προκειμένου να αποτεχτούμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τους υπόλοιπους ε, σκιώδεις. Η Κάρεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ εισηγητά για την ε, παρουσίαση αυτή. Για τα δημοσιονομικά μακροπρόθεσμα και για τη βιώσιμη διαμόρφωσή τους, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται και σε βραχυπρόθεσμο πλαίσιο. Θεωρώ ότι καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ανεύθυνο να μεταφέρονται τεράστια δημόσια χρέη στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι πραγματικά ανεύθυνο σε περιόδους τέτοια τεράστια γύρανσης του πληθυσμού, όπου θα αυξηθούν οι πιέσεις. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα διαφορετικό σημείο κίνηση σε σχέση με τον εισηγητή μας. Φυσικά τα σωστά δημοσιονομικά είναι πάρα πολύ σημαντικά για, την, ε, για τον περιορισμό της, ε, του πληθωρισμού αλλά βλέπω ότι ο εισηγητής αναφέρεται σε θέματα ανάπτυξης. Αλλά υπερβάλλει. Με το κριτήριο της ε, πλήρους ε, ανάπτυξης του δυναμικού παραγωγής, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι, Πρόεδρε, δεν είναι σωστός αυτός ο δρόμος. Έχουμε ένα πακέτο ανάπτυξης και τι μας καταδεικνύουν τα τελευταία χρόνια, ότι στις καλές εποχές ίσως δεν τηρούνται επαρκώς τα κριτήρια του Συμφώνου σταθερότητα και γι' αυτό σήμερα καταλήγουμε σε τόσο προβληματικές καταστάσεις. Θα πρέπει να έχουν τηρηθεί πιο αυστηρά τα κριτήρια αυτή και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, ε, συγγνώμη, ευρωπαϊκή διακυβέρνηση σε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πειθαρχία και έλεγχος σε αυτή την, ε, από αυτή την ε, άποψη. Τη στιγμή που η Γερμανία και η Γαλλία, οι μεγάλες χώρες αυτές, ε, μιλούν για ευελιξία, δεν τηρούνται επαρκώς τα κριτήρια αυτά. Κάτι άλλο Νομίζω ότι αυτό που προδιαγράφεται προϋποθέτει ένα ευρωπαϊκό κεντρικό κράτος και δεν ε, επιτρέπει αρκετές ε, αρκετή επικοινομορφία. Εγώ υποστηρίζω την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις συντάξεις και αυτό είναι δυνατόν εάν τηρηθούν και εποπτεύονται πιο αυστηρά τα κριτήρια σταθερότητας προκειμένου να μην έχουν τόσο μεγάλο περιθώριο ελιγμού τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα αυτό να αποτελέσει το βασικό στοιχείο στην έκθεσή σας όλοι. Ο Ούντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαι απόλυτα βεβαίω για το εξή. Αν ε, υπήρχαν πιο πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ε, εδώ στην αίθουσα και άκουγαν αυτά που είπε ο συνάδελφος Νόκ, θα ανησυχούσαν ακόμα πιο πολύ από τη σήμερα, γιατί μέχρι αυτή τη συζήτηση θεωρούσα ότι εμείς στην Επιτροπή κάτι είχαμε διδαχθεί από την όλη κρίση, από την όλη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Θεωρούσα ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια σωστή συζήτηση για το τι θα πρέπει να αποτελέσουν, από τι θα πρέπει να αποτελείται η δημόσια δράση. Και είχα την εντύπωση ότι ο λαϊκισμός όπως είπε ο κύριος Χόικμαρκ, δεν είναι όπως παλιά. Δεν μπορεί στα σοβαρά κανείς να πιστεύει ότι όταν το τριπλάσιο του ΑΕΠ της Γερμανίας, της πιο σημαντικής και μεγάλης δημοκρατίας ε, οικονομίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει χαθεί. Αυτό έχει να κάνει με τις προτάσεις που έγιναν εδώ πέρα τις ε, τελευταία χρόνια. Πόσο μπορεί κανείς να απέχει από την πραγματικότητα για να ε, εκφράσει αυτή την ιδέα και δεν θα πρέπει να ξεκινήσει διάφορες λαϊκιστικές διακήρυξεις ο κύριος ε, από τους πράσινους. Γιατί αυτό που απασχολεί πραγματικά τον κόσμο είναι πόση καινούρια, πόση νέα ε, κοινωνική ένδια θα προκύψει. Πόσοι θα πληχθούν ακόμα. Και συμφωνώ με τη συνάδελφο Βόρτμαν Κόλ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμασταν αρκετά αυστηροί με τους όρους που θέσαμε στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Όχι, δεν ήμασταν αρκετά έξυπνοι, αν θέλετε. Δεν ήμασταν αρκετά έξυπνοι, γιατί δεν προσπαθήσαμε να επενδύσουμε εκεί όπου ήταν σημαντικό και λογικό να επενδύσουμε για να οικοδομήσουμε μια νέα οικονομία. Όχι. Αυτό ήταν, ε, εκεί αποτύχαμε. Και κανείς δεν θα εξέλθει από την οικονομική αυτή κατάσταση ακολουθώντας απλά ιδεολογίες. Είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό. Και με τη συζήτηση αυτή δεν πρόκειται να συμβάλλουμε επουδενή στην επίλυση της κατάστασης. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα βγούμε από την παγίδα των χρέων. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μέσω της ανάπτυξης. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό ε, προσπαθώντας να καταστρέψουμε με οικονομίες, με περικοπές Τη ευρωπαϊκές οικονομίες. Και γι' αυτό πρέπει να πω στον συνάδελφο Γκίγολτ ότι είμαστε ανοιχτοί για μια σωστή συζήτηση για το πώς θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί η βιομηχανία και η οικονομία. Αυτό είναι σημαντικό και σίγουρα θα αποτελέσει και το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων μας. Μπορούμε λοιπόν να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε την περαιτέρω αποδυνάμωση του κράτους για την περαιτέρω ε, έκρηξη, αν θέλετε, και αύξηση της ανεργίας. Δεν είναι δυνατόν έτσι να ελπίζουμε ότι θα βγούμε από την κρίση, ότι θα βγουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες από, από την κρίση. Θα πρέπει να βρούμε λογικές νέες λύσεις και να μην πέσουμε πάλι στις παλιές ιδεολογικές παγίδες, γιατί δεν μας βοηθούν καθόλου. Uh, right. Kate Swinburne. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από τους ε, που ε, με άκουσαν ήδη να λέω αυτή τη βδομάδα τα ίδια πράγματα ότι μιλάμε για ε, την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας ε, ανησυχώ. Μήπως δεν έχουμε καταλήξει σε ένα σωστό ορισμό του δημοσίου χρεούς. Μετά το ΕΚΟΦΗΝ της περασμένης εβδομάδας προέκυψε σαφώς ότι ούτε εκείνοι ξέρουν ακριβώς πώς να ορίσουν το δημόσιο χρέο. Μέχρι να βρούμε κριτήρια λοιπόν σχετικά με το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και τι όχι, κυρίως όταν μιλάμε για τον ισολογισμό, θα δούμε ότι πολλά κράτη-μέλη χρησιμοποιούν πολλά τέτοια χρηματοπιστωτικά εργαλεία του ισολογισμού ε, και θα τα συζητήσουμε αυτά όταν πιάσουμε το θέμα των παραγόγων, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις, ε, συνταξιδοτικές υποχρεώσεις ε, που ε, δεν έχουν την επαρκή χρηματοδότηση. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται με τον ισολογισμό και να ορίζουμε επακριβώς το δημόσιο χρέος. Κάτι άλλο πρέπει να προσέξουμε στη συζήτησή μας ε, είναι ότι ε, τα κράτη-μέλη δανείζονται από τους επενδυτές ε, μέσω των αγορών και ε, χρειάζονται ποσά άνευ προηγουμένου. 30 δις χρειάζεται η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία και την Πορτογαλία που κάνουν rollover που αντιστοιχεί σε 20-27% του ΑΕΠ τους. Για ευρωπαϊκά δεδομένα είναι υπέρογκα αυτά τα ποσά. Οπότε χρειαζόμαστε μια στρατηγική ώστε όταν απευθύνονται στις αγορές για να δανειστούν τα κράτη θα πρέπει να το έχουν υπόψη αν υπάρχει δηλαδή επιλογή ανάμεσα στα, στις χώρες της ζώνης ευρώ Υπάρχει πληθώρα επενδυτών. Δηλαδή, θέλετε να, το χρέος της Γερμανίας ή κάποιας άλλης ε, χώρας και, υπάρχει και υπάρχουν και χώρες εκτός ζώνης ευρώ. Η καποιας αλλης χωρας και και υπαρχουν και χωρες εκτος ζωνης ευρω η χρηση των ε, παραγόγων ε, δεν μας δείχνει ότι πολλά ομόλογα ευρώ μετατρέπονται σε άλλα νομίσματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σωστοί ορισμοί και να προσέξουμε απλά πράγματα, έστω και βραχυπρόθεσμα, ώστε να μην έχουμε κρίση και με τα κρατικά χρέη, πέρα από την κρίση των δημοσιοοικονομικών. Ευχαριστούμε. Κυρία Γιαζοβιέσκα, επιστρέψατε παρακαλώ. Έπρεπε να πάω στην Επιτροπή, να μεταβώ στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, θα ήθελα να σας πω λοιπόν, καταρχήν, σε σχέση με την έκθεση του κ. Γκόκ ότι θα πρέπει να δούμε ορισμένες πτυχές οι οποίες δεν ε, λήφθησαν υπόψη και είναι πολύ σημαντικές. Η στρατηγική εξόδου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ορίσουμε τις ε, προτεραιότητες της μακροχρόνιας επένδυσης που θα αποδώσουν μακροχρόνια ως προς την οικονομική ανάκαμψη. Άρα η πρωταρχική επένδυση θα πρέπει να γίνει στην έρευνα και ανάπτυξη, στην κατάρτιση και στην ε, ενδυνάμει ανάπτυξη. Στην αγορά εργασία. σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι τόσο κινητικοί και δημιουργική ή άλλοι που μπορούν να ανταποκριθούν με ευελιξία στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να επισύρουμε την προσοχή στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν, να ληφθούν σημαντικά μέτρα υπέρ της οικονομίας της αγοράς και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλοι οι πόροι και το ε, ανθρώπινο κεφάλαιο, το έμψυχο υλικό. Να δούμε και την ε, μετανάστευση, διότι οι μετανάστες, οι μετανάστες δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα κενά στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να σταθούμε στα προγράμματα υπέρ των εργαζομένων άνω των 50 καθώς και υπέρ των νέων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τα συνταξιοδοτικά. Τώρα, ως προς τη μακροχρόνια σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές, την κοινωνία που γυράσκει, Λουένα και γυράσκει. Θα πρέπει να δούμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, Βλέπουμε ότι οι δημογραφικές αλλαγές, ο αντίκτυπος τους έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με την τρέχουσα κρίση. Νομίζω ότι έχει σημασία για τα δημοσιοοικονομικά, διότι οι μεταγενέστερες γενές θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Η κυρία Κόλτο ανέφερε αυτό. Η φορολογική πολιτική θα πρέπει να οδηγήσει σε μία εξισορρόπηση μεταξύ γενεών. Και αυτό μέσα στα πλαίσια της ε, σταθερότητας της μακροχρόνιας πολιτικής. Τώρα, στην τρίτη παράγραφο, πώς αναγνωρίζουμε το δημόσιο χρέας, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία εποπτεία και του συνταξιοδοτικού και να μην μιλάμε για τις υποχρεωτικές δαπάνες του δημόσιου τομέα, αλλά εν γέννη τον δημόσιο τομέα, ο οποίος θα ορίσει καλύτερα τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Eurostat θα πρέπει να ορίσουν μια κοινή μεθοδολογία για τέτοιες εκθέσεις. Επίσης, όπως ε, όσον αφορά τη διαχείριση της φερεγγιότητας, Νομίζω ότι οι ολοένα και μεγαλύτερες αλλαγές μειώνουν το κόστος ε, ε, εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τη ρευστότητα και τη φερεγγιότητα ως προς τα δημόσια οικονομικά. Όταν μιλάμε για επανακαταβολές των κρατικών επιχορηγήσεων, ιδιαίτερα για χώρες με υψηλό έλλειμμα. Δεν μιλάμε μόνο για καλύτερη διακυβέρνηση, για περισσότερες υπηρεσίες IT. Πολλές φορές το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό και εδώ μπορούμε να μειώσουμε το κόστος, τουλάχιστον βραχυκρόθεσμα. Ο Ζαν Πολ Γκοζές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του. Ε, τουλάχιστον υπάρχει ένα αξιόλογο στοιχείο. Προσπαθεί να εχνηλατήσει ορισμένες ε, ενδεχόμενες λύσεις, η επιλύση του ζητήματος. Διότι, όπως είπε ο Ούντο, και επειδή εγώ είμαι ένας ε, πολίτης, δήμαρχος μιας, ενός μικρού χωριού, μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν ε, μας οδηγούν σε λύση. Όταν μιλάμε για μείωση των δημόσιων δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι μειώνουμε τα εισοδήματα και για μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε το θάρρος να πούμε ότι αυτό σημαίνει αυστηρά δημόσια οικονομικά, άρα θα πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι. Όλοι. Στην Γαλλία υπήρξε μια πρημοδότηση για την απόσυρση των αυτοκινήτων. Πολύ καλή ιδέα, διότι έτσι αγοράστηκαν πολλά καινούργια αυτοκίνητα και εκείνοι που ασχολούνται με τον τεχνικό έλεγχο των μεταχειρισμένων τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, διότι τα νέα αυτοκίνητα δεν, δεν υφίστανται τον έλεγχο των κταίων τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια, άρα μειώνεται το τζίρος τους. Οι καθηγητές ε, μακροοικονομικών θα το τόνιζαν αυτό. Όλα είναι αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δηλαδή κάτι αντιστοιχεί σε κάτι άλλο. Μιλάμε για μία εύθραυστη ισορροπία στις οικονομίες μας και ιδιαίτερα στις προηγμένες οικονομίες και αν πέσει ένα κομμάτι του ντόμινο θα πέσουν όλα. Μιλάμε για χρηματοδότηση εκπαίδευση, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχει όμως μεγάλο χάσμα μεταξύ της ποιότητα εκπαίδευση και των αναγκών της οικονομίας. Η κατάρτιση δεν αντιμετωπίζεται σωστά, τουλάχιστον στη χώρα μου, και δεν υπάρχει σωστή αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης. Ε, μιλάμε για το συντοξιοδοτικό μπορούμε να προωθήσουμε το συνταξιοδοτικό τουλάχιστον σε σχέση με μία ε, ισότιμη βάση χωρίς να, να θίξουμε το όλο οικοδόμημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες ε, ότι βγάζουμε τα χρήματα από τον ένα τομέα για να τα βάλουμε κάπου αλλού. Μειώνουμε κάτι για να αυξήσουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν αυτές δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε πραγματιστές. Αμφισβητούμε πολλά στοιχεία, αλλά τουλάχιστον η έκθεση προσπαθεί να βάλει τα πράγματα κάπως στη θέση τους. Και εμείς με τις τροπολογίες μας προσπαθούμε να δώσουμε σωστές αποχρώσεις. Γιατί πώς μπορούμε να μιλάμε για δημόσια οικονομικά που να έχουν εξηγιανθεί τη στιγμή που δεν υπερβαίνουμε τα δύο χρόνια απασχολησιμότητας. Ε, βλέπουμε στη Δημαρχία ότι έχουμε προγράμματα εξοπλισμών τα οποία δυστυχώς ε, δεν, έχουν, ε, δεν μπορούν να ζήσουν για πολλά χρόνια. Εμείς κάνουμε πλατείες με λουλουδάκια αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Οι δημόσιες πλατείες δηλαδή με τα λουλουδάκια τους. Έντουαρντ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή με τη σειρά μου για αυτή την έκθεση. Δεν θέλω να μιλήσω για τις λύσεις όπως οι συνάδελφοι. Θα ήθελα μάλλον ε, να μιλήσω για τις εκθέσεις, ε, για την υποβολή αναφορών. Γιατί τι να τις κάνουμε τις δομές και τις λύσεις για με ένα τέτοιο σύμφωνο ε, απο... Ε, ενώ δεν ακολουθείται δημοσιονομική πειθαρχία από τα κράτη-μέλη για τη μέτρηση ε, του χρέους, της προβλέψεις του ΑΕΠ, ό,τι και να μετρούν. Και μετά περνάει στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και στις αγορές γενικότερα. Για τα κριτήρια του Μάστριχτ το ίδιο είναι. Υπάρχουν τα κριτήρια, καλά είναι. Αλλά είδαμε πρόσφατα τι συμβαίνει όταν ένα κράτος ε, μέλος δεν ε, κάνει πιστή απογραφή των στοιχείων εις βάρος των υπολείπων. Τώρα όταν μιλάμε για δημιουργική λογιστική, όπως θέλετε πείτε το, τελικά είναι ένα απαρχαιωμένο λογιστικό ε, σύστημα. Πώς γίνεται χώρα της Ευρωζώνης ε, τώρα να κάνει τους λογαριασμούς της σε βάση των μετρητών, ενώ όλα εξαρτώνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Δηλαδή θα κρατήσει τις επιταγές ε, που στο σιρτάρι, τις επιταγές με τα χρήματα που πρέπει να καταβληθούν σε διάφορους φορείς του δημοσίου. Δική του η επιλογή δεν πρέπει να επιτρέπεται αυτό στο μέλλον ε, θα πρέπει η Επιτροπή να έχει το, τη δυνατότητα ελέγχου, στενή παρακολούθηση και των αποτελεσμάτων και των προβλέψεων. Γιατί οι προβλέψει ε, δεν είναι ακριβή επιστήμη, αλλά άλλο μια πρόβλεψη με μικρά λάθη και άλλο ε, μια πάντοτε αισιόδοξη πρόβλεψη, ούτω ώστε να δίνετε την εντύπωση ότι πρόβλημα δεν υπάρχει και ότι έχετε έτοιμη την λύση. Ε, ε, ε, υπερεκτιμώντας το ΑΕΠ Στην έκθεση θα ήθελα να αναφερθούμε στην διαχείριση των στατιστικών Ινστιτούτων για ανεξάρτητα στατιστικά ιδρύματα, ε, για εκθέσεις σχετικά με τις συντάξεις, ΑΕΠ, ε, για σαφή ακριβή μέτρηση, για τα δεδομένα που είναι σημαντικά και συμβάλλουν στο να εξευρεθούν οι λύσεις που σήμερα συζητούμε. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ να πω κάποια πράγματα. Πρώτον, μία εξαγγελία. Αυτή η έκθεση γίνεται σε ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης. Και η Επιτροπή Απασχόλησης ε, θα ε, εστιαστεί στις στρατηγικές εξόδου και τις ε, κοινωνικές διαστάσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές και μεριμνώντα, ούτω ώστε τα συστήματα κοινωνική ασφάλισης να είναι βιώσιμα. Όλα αυτά τα ζητήματα που προανέφερα είναι μάλλον αρμοδιότητα τη επιτροπή απασχόληση και άρα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με εμά. Ε, θα υπάρχουν δύο μέρη σε αυτή την έκθεση, δύο εκθέσει συγχωνευμένε, αν θέλετε. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας λέω να μην μπαίνετε, στα χωράφια της Επιτροπής Απασχόλησης γιατί όλα τα στοιχεία είναι αλληλένδετα. Εφιστώ είναι προσοχή σας πάντως ότι στο μέτρο του δυνατού πρέπει να προσπαθήσετε να ασχοληθείτε με ζητήματα που εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα. Και η Κέιτ και ο Έντουαρτ κρίνουν ότι έκαναν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με την παρακολούθηση, δηλαδή τι συμπεριλαμβάνει τελικά το έλλειμμα. Ε, σαφώς Έχουμε φτάσει στο σημείο που χρειαζόμαστε νέα εργαλεία για να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε καλύτερα τι έχουν συμπεριλάβει στους λογαριασμούς τους τα κράτη-μέλη. Στην ακρόαση για τον νέο Επιτροπό Λιρέν, ε, το θέμα της λογιστικής καταγραφής εκτός ισολογισμού αναφέρθηκε και του ζητήσαμε να το ε, διερευνήσει και μετά η Κέιτ έκανε περώτηση και είπε ο κύριος Όλη θα το διερευνήσει. Ε, βέβαια έχουν έκτοτε σημειωθεί εξελέξεις, πάντως ε, στον τύπο είπα ότι ασχολείται με το ζήτημα το Κοινοβούλιο και ότι όντως χρήζει διερεύνησης ε, το θέμα αυτό. Αύριο κάνουμε ανταλλαγή απόψεων για την πρώτη έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Στατιστική Διακυβέρνηση. Έχει σημασία και σε αυτό το θέμα όχι επειδή ήμουνα εγώ που συγκρότησα τη Συμβουλευτική Επιτροπή και αγωνίστηκα για να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη για οποιοδήποτε είδους αλληλοεπιτήρηση των στατιστικών στοιχείων, αλλά είναι σημαντικό να προχωρήσουμε και γι' αυτό και για άλλα ζητήματα. Έχουμε την ευκαιρία τώρα να ανοίξουμε περισσότερο την πόρτα ε, και να υπάρξει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Σκεφτείτε το και αυτό. Ε, είπα ότι χρειαζόμαστε εργαλεία παρακολούθησης ε, και δεν είμαστε σίγουροι ότι συμπεριλαμβάνεται στο έλλειμμα, αλλά ε, δεν δικαιολογεί αυτό την αργή πρόοδο. Όσο και να είναι το έλλειμμα, σε κάθε περίπτωση μεγάλο είναι αλλά υπάρχει και ανάκαμψη, υπάρχει το θέμα του χρονισμού των δράσεών μας. Ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει πάντως τα απαιτούμενα εργαλεία για μια επακριβέστερη παρακολούθηση των στοιχείων και δεν κατανοούμε ακριβώς όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο, στο έλλειμμα, αλλά δεν μπορούμε αυτό να το προτάξουμε ως ε, λόγο για να εγκαταλείψουμε το θέμα των ελλημάτων. Ο κύριος Βάης είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θα θέλατε να σχολιάσετε αυτό το ζήτημα. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με τις ε, προτάσεις οι οποίες ε, αναφέρονται στην έκθεση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάγκη για μεγαλύτερο στατιστικό ορθολογισμό, καλύτερους δείκτες, καλύτερους ορισμούς. Και ασφαλώς και όλα αυτά θα τοποθετηθούν στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασίας. Ωστόσο, έχουμε κάποιες αμφιβολίες επί της έκθεσης που αποστέλνει κάποια μηνύματα τα οποία ενδεχομένω να παρερμηνευτούν. Να αναφερθώ σε ορισμένα εξ αυτών. Καταρχάς, Πιστεύουμε ότι η έκθεση βασίζεται σε μια στενή θεώρηση του ρόλου των δημοσιονομικών. Ενώ η πολιτική, η αντικυκλική αποτελεί σημαντική δύναμη στην πολιτική ανάπτυξη, οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν καταδείξει ότι τίθενται πολλά θέματα λόγω αναγκών προσαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες με μεγάλες ε, εξωτερικές και εσωτερικές αστάθειες θα πρέπει να προσαρμόσουν ε, την αντιμετώπιση τους ανάλογα με τον αντικυκλικό τους αυτό, την αντικυκλική φάση. Κατά δεύτερον, ε, η έκθεση που ανέφεραν πολλοί ομιλητές δεν δημιουργεί, αν θέλετε, απαραίτητα την σχέση μεταξύ βιωσιμότητας και της γύρανσης. Ακόμα και πριν από την κρίση οι πρακτικές ήταν μη βιώσιμες και χρειαζόταν αποφασιστική δράση για να μην ε, εκραγούν τα χρέη. Η κρίση υπογράμμισε, απλά τόνισε αν θέλετε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να επανέλθουμε σε βιώσιμο επίπεδο τα δημοσιονομικά. Κατά τρίτον, η ανάγκη διορθωτικών μεταρρυθμίσεων για την αύξηση της ανάπτυξης είναι σημαντική και θα πρέπει προφανώς να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα αυτό. Ωστόσο, έχουμε κάποιες αμφιβολίες για τις προτάσεις που κάνει ο εισηγητής σε ό,τι αφορά περιπτώσεις κακοδιαχείρισης. Γι' αυτό λοιπόν θα προτείναμε να βελτιωθεί η έκθεση, να δοθεί πιο ευρία θεώρηση σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να καταλήξουμε σε βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική. Αυτό καταρχάς σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις χρηματοοικονομικές ε, προσπάθειες που προτείνονται και θα πρέπει να ξεκινήσει σε πολλές ε, χώρες ε, ένας εξοχρολογισμός σε ό,τι αφορά τις προσαρμογές που είναι απαραίτητες σε κάποιες χώρες οι οποίε θα πρέπει να, ξε... ξεκινήσουν τώρα. Οι μεταρρυθμίσει τώρα στο κοινωνικό σύστημα, στο σύστημα δεξιοδότηση και το σύστημα υγειονομική περιθέψη θα πρέπει να προσαρμοστούν στα δημοσιονομικά και θα πρέπει να γίνουν διαχρονικές μεταρρυθμίσεις για να προωθηθούν οι επενδύσεις θεωρούμε ότι αν συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία στην έκθεση, θα δοθεί μια πιο ευρεία προοπτική στην όλη έκθεση, η οποία είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο εισηγητή θέλει να κλείσει τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια και μόνο. Το εγχείρημα ήταν πολύ σημαντικό. Ενείχε πολλά στοιχεία, άρα δεν μπορούσα να τα συμπεριλάβω όλα. Γιατί στις διάφορες παρεμβάσεις μου ζητήσατε να αντιμετωπίσω και διάφορα επιμέρους ζητήματα. Στη συνέχεια ήμουνα πολύ συνετός, διότι θεώρησα το σύμφωνο σταθερότητας αποτελεί δέσμευση με βάση την αναθεώρηση του 2007 και ε, όρισα το δεσμευτικό πλαίσιο των συνθήκων και των κοινοτικών κειμένων. Σε αντίθεση με άλλες εκθέσεις όπου ορισμένοι συνάδελφοι μιλάνε για τη χρηματοδότηση του δημόσιου ελλείμματος μέσω ευρωμολόγων, κάτι που απαγορεύει η συνθήκη της Λισαβόνας, ή την χρηματοδότηση του δημοσίου ελλείμματος κάνοντας αυτό που κάνανε οι ΙΠΑ, δηλαδή να επιτεθεί, να επιτεθεί κερδοσκοπικά κατά της Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας. Δηλαδή με μηδενικό επιτόκιο, να επιτεθεί με μηδενικό επιτόκιο. Εγώ δεν έλαβα υπόψη αυτό το στοιχείο. Παρέμενα λοιπόν μέσα στα πλαίσια των κοινοτικών και συμβατικών δεσμεύσεων και προσπαθώ σε αυτή την ε, έκθεση να προωθήσω ένα διάλογο μεταξύ μας για να φτάσουμε σε έναν κοινό παραγνωμαστή, παραγνωμαστή δηλαδή την υποστήριξη των δημοσίων οικονομικών. Και αρκέστηκα σε αυτό. Σε σχέση με αυτό το εγχείρημα, και εγώ ανησυχώ συνάδελφοι, και αυτό το λέω και στους συντηρητικούς και στους ε, φιλελεύθερους. Εάν δείτε εκ του σύνεγγης την εξέλιξη της διάρθρωσης των προϋπολογισμών στα κράτη-μέλη μας, τι παρατηρείτε. Παρατηρείτε ότι το μέρος, το μερίδιο των δημόσιων δαπανών στο ΕΠ δεν έχει αυξηθεί και σε ορισμένες χώρες έχει μειωθεί. Και το θέμα του ελλείμματος οφείλεται, και μιλώ για την πρόσφατη περίοδο, στην ε, μείωση των δημόσιων εσόδων. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί και γι' αυτό ανησυχώ και απευθύνομαι στην Επιτροπή. Με ενδιαφέρει λοιπόν η αποτελεσματικότητα των δημόσιων οικονομικών και του φορολογικού πλαισίου που ίσχυσε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζοντας την οικονομία μέσω της προσφοράς. Δηλαδή οι δημόσιες δαπάνες τι έχουν κάνει, έχουν ακροτηριώσει τον προϋπολογισμό. Μέσα στα πλαίσια ενός αυστηρού πλαισίου, χωρίς να υπάρχουν προοπτικές ως προς την ανάπτυξη, εάν μειώσετε τους φόρους, για παράδειγμα, και έχετε έναν αναπτυξιακό στόχο 2% και η οικονομία βρίσκεται κάτω από αυτό το 2% τι γίνεται. Αυτό το έλλειμμα ολοένα και βαθαίνει, όχι μόνο γιατί αυξήσατε τις δημόσιες δαπάνες, αλλά γιατί μειώσετε και την φορολόγηση και η ε, μείωση της φορολόγησης δεν οδηγεί σε ε, αναπτυξιακή πορεία υποχρεωτικά. Άρα ε, κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα. Και αυτή είναι και η πρωταρχική μου ανησυχία, δηλαδή η μη αποτελεσματικότητα των φορολογικών δαπανών. Άρα ανησυχώ όσο και εσείς για αυτή την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, διότι οι δημόσιες δαπάνες στις περισσότερες χώρες έχουν παραμείνει στις, στις περισσότερες χώρες σε επίπεδο πριν της ε, κρίσης, στο πρώτης κρίσης επίπεδο. Άρα αν σήμερα περικόψουμε τις ε, δημόσιες δαπάνες και ιδιαίτερα τις ε, κοινωνικές δαπάνες σε αντίθεση με τους στόχους μας, στην ουσία ε, μεγαλώνουμε το έλλειμμα. Άρα δεν υπάρχει ανάκαμψη, διότι εάν στοιχηματίσουμε και αν όλες οι χώρες ακολουθήσουν μια πολιτική αυστηρότητας με από πληθωρισμό στους μυθούς δεν θα υπάρξει αναπτυξιακή πορεία. Και αυτό αφορά τις δημόσιες δαπάνες, διότι ε, δυστυχώς η ύφεση, η ύφεση θα επανέλθει. Και πιστεύω ότι τα προσδοκόμενα αποτελέσματα δεν θα ισχύσουν. Και εδώ βλέπετε ότι η κερδοσκοπία των αγορών θα πλήξει ακόμα περισσότερο την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτοκαλία. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε και γι' αυτό σήμερα πρέπει να διανοίξουμε μια νέα οδό. Γι' αυτό μίλησα για την υποστηριξιμότητα των δημοσίων δαπανών μακροχρόνια. Υπάρχει μια σειρά προτάσεων θα τις μελετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν θέλουμε να αυξήσουμε το έλλειμμα. Στο τέλος της δεκαετίας του 80, όταν βρισκόμασταν σχεδόν στην πλήρη απασχόληση, εμείς, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, θα έπρεπε τα έσοδα αυτά, αυτού του φορολογικού καλαθιού, θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε το χρέος μας. Και αυτό αφορά το φορολογικό. Βλέπετε ότι είμαι αρκετά ορθόδοξος. Σε σχέση με την πλήρη απασχολησιμότητα θα πρέπει να έχουμε μία, έναν, ισολο, έναν σωστό ισολογισμό. Αλλά τη στιγμή που έχουμε τόσο υψηλό επίπεδο ανεργίας, το υψηλότερο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο αυστηρό πλαίσιο δημοσίων οικονομικών. Θα πρέπει να έχουμε μία εξισορρόπηση, ένα πάγωμα δηλαδή για τρία με πέντε χρόνια. Ως προς τις συντάξεις, μου υποβάλλατε ένα ερώτημα για το συνταξιοδοτικό. Δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση, πώς θα διαμορφωθεί για το 2050. Αυτός ο οποίος μπορεί να ορίσει τα δημογραφικά μας το 2050, το δίκτυο γονιμότητας, ε, ποιο τμήμα των μισθών θα ορίζει το συνταξιοδοτικό πώς θα έχει η μεταναστευτική ροή, μπράβο, εγώ δεν μπορώ. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην δραματοποιούμε. Στην αιτιολογική σκέψη σας δίνω αυτά τα στοιχεία, δεν τα αγνώ, αλλά όπως ε, υπενθύμησε και η Πρόεδρος, θα πρέπει να γίνει ένας επιμερισμός εργασίας σε αυτή την έκθεση. Θα πρέπει η Επιτροπή Απασχόλησης να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα και εγώ αρκέστηκα να υπενθυμίσω και να πω ότι αν το κοινωνικό μοντέλο είχε μία χρησιμότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης, τότε η Επιτροπή Απασχόλησης θα έπρεπε να εξεύρει τις κατάλληλες λύσεις για την ε, διαιώνιση αυτού του μοντέλου. Εγώ προσπάθησα να βρω δείκτες που να αρμόζουν σε όλους. Σε σχέση με τον ενδυνάμει δείκτη ανάπτυξης και την ε, δυνατότητα χρήσης, ε, πραγματικής χρήσης της παραγωγής. Οι οικονομολόγοι θα θέλουν να ξέρουν ποιος είναι ο δείκτης ανάπτυξης σε κατάσταση πλήρους απασχόληση δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες παραγωγής, κάτι το οποίο θα ήταν κατόφλι για να φτάσουμε σε μια πολιτική εξόδου μέσα στα πλαίσια των διαρθρωτικών πολιτικών που ορίζει η Επιτροπή. Η Επιτροπή πιστεύει ότι εν δυνάμει δείκτης ανάπτυξης της Ευρώπης έχει μειωθεί σε 1-1,5%, γι' αυτό θα πρέπει να εξεύρουμε πολιτικές εξόδου. Εάν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αν και θεωρώ ότι ο ενδυνάμει δείκτης ανάπτυξης ίσως υπερβαίνει το 1,5%. Γι' αυτό χρειάζεται υποστήριξη με σταθεροποιητές. Αλλά για να ξεφύγουμε από αυτή την τρελή συζήτηση, εγώ πήρα τον δείκτη που λαμβάνουν υπόψη όλοι οι οικονομολόγοι, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη εν δυνάμει χρήσης της παραγωγής. Εδώ βλέπουμε ότι οι μηχανές κινούνται κατά 70%, δηλαδή η ε, παραγωγιμότητα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς κινείται αυτός ο μηχανισμός να βρούμε δηλαδή ε, ενέργειες έφνης που να μην ε, μολύνουν. Εγώ προτείνω την ίδια λογική να χρησιμοποιήσουμε και εδώ, αλλά δεν εξαντλούμε την όλη συζήτηση ως προς το επίπεδο ε, επένδυσης. Αναμένω λοιπόν υποδείξει από τους πρασίνους που είναι και οι πλέον αρμόδιοι. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστηκε η συζήτηση γιατί ε, αναβλήθηκε η έκθεση Λάγκεν και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε πιο διεξοδικά. Η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 5η Μαρτίου και να λάβετε υπόψη ότι στις 3 Μαρτίου αναμένουμε τις προτάσεις Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Αν θέλετε να τις λάβετε υπόψη στις 22 Μαρτίου θα δούμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 27 Απριλίου. Άρα έχουμε αρκετό χρόνο για διαπραγματεύσεις. Και στην Ολομέλεια του Μαΐου 2 θα δούμε την έκθεση και θα είναι έτοιμη για τον Ιούνιο, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα μέχρι τότε, αλλά θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ουσιοδός. Τελικό θέμα στη σημερινή ημερήσια διάταξη είναι το 8 σε σχέση με το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιριών και ούτω καθεξής. Κύριος Καντράουε, ευχαριστώ Πρόεδρε και καταρχά, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονό ότι είναι δύσκολη η χρονική συγκυρία για μένα γιατί θα πρέπει να προσιάσω μια άλλη έκθεση σε άλλη επιτροπή λίγο μετά τι 5. Ανακοίνωσα ωστόσο ότι θα καθυστερήσω λίγο. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Συνάδελφοι θα θυμάστε τις συστάσεις της Επιτροπής ε, τέλη Απριλίου 2009 σε ό,τι αφορά τις αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, σε ό,τι αφορά δηλαδή συγκεκριμένα και τις συγκεκριμένες εταιρείε. Και αυτές οι συστάσεις θα αποτελούν τη βάση των εργασιών μου και των προτάσεών μου. Αλλά ήδη γίνονται και έχουν λεφτεί διάφορες πρωτοβουλίες σε διάφορα φόρα και υπάρχουν και πολλές εθνικές πρωτοβουλίες. Είναι σημαντικό λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαμορφώσουμε μια αποκρισταλωμένη ε, και σωστή, ολοκληρωμένη άποψη. Ε, λόγω της οικονομικής κρίσης ε, Υπόκειται μεγάλη πίεση φυσικά και οι εταιρείε και οι τράπεζε. Αυτό αποτελεί την ηθική πτυχή. Αλλά θα πρέπει να πούμε επίση ότι ο οικονομικό αντίκτυπο τη πολιτική αυτή και η υπερβολική εστίαση στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο συμβάλλουν ασφαλώς ε, στο βάθος της ε, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται μεγαλύτερη τυποποίηση, μεγαλύτερη ρύθμιση και επαναλαμβάνεται αυτή η ανάγκη. Η πιο καλή ρύθμιση της πολιτικής των αποδοχών θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θεωρώ, σε ό,τι αφορά τις κεφλακίες απαιτήσει, την εποπτεία και η συνάδελφος Μακάρθη θα ασχοληθεί στην έκθεση της ε, με τα θέματα αυτά. Η δική μου έκθεση εστιάζεται πιο πολύ στις γενικές αρχές προκειμένου να διαμορφωθεί μια βέλτιστη πολιτική αποδοχών σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές εταιρείες, τις, τράπεζες αλλά και τις συγμένες εταιρείες. Και θα πρέπει να σκεφτούμε σε ποιο βαθμό οι συστάσεις ε, αυτές θα πρέπει να καταστούν πιο ε, δεσμευτικές, γιατί ε, έχει καταδεχτεί ότι δεν επαρκούν απαραίτητα οι συστάσεις για να δημιουργηθεί ίσο επίπεδο ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελέτες και οι μελέτες του τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αναφέρουν κάποιες συγκεκριμένες τάσεις, για παράδειγμα μεταξύ συνδέσμου και σύνδεσης ε, της κακής κατάστασης ε, της οικονομίας και της πολιτικής αποδοχών. Και τι διαπιστώνουμε, ότι καταρχάς τα τελευταία 15 χρόνια υπήρξε μεγάλη αύξηση της, των μέσων αποδοχών των διευθυντών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αύξηση του μεταβλητού στοιχείου των αποδοχών. Κατά δεύτερον, οι αναλύσεις καταδεικνύουν ότι υπάρχει ε, ανεπαρκής σύνδεση μεταξύ των, ε, της αύξησης των αποδοχών των διευθυντικών στελεχών και της γενικότερης απόδοσης της εταιρεία. Αυτά προκύπτουν και από τη γενική από τον Παγκόσμιο Οργανισμό εργασία Κατά το τρίτον, βλέπουμε ότι είναι πολύ υψηλό το μεταβλητό στοιχείο αυτό κατά μέσο όρο. Και από δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι δεν ε, διστάζουν να κάνουν περικοπές στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Με άλλα λόγια δηλαδή, ότι υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο, μια βραχυπρόθεσμη διάσταση και παράλληλα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουν ληφθεί ε, και διάφορες εθνικές πρωτοβουλίες για να υπάρξει καλύτερη σύνδεση μεταξύ των αποδοχών και της απόδοσης των CEOs, των διευθυντικών στελεχών. Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία έχουν ληφθεί έχουν λάβει τέτοιες ε, πρωτοβουλίες, αλλά πέρα από τις ε, πρωτοβουλίες αυτές. Υπάρχουν φυσικά διαφορές σε ό,τι αφορά τη φορολογική πολιτική, στην εταιρική πολιτική και όλα αυτά. Και άρα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει έτσι εύκολα και γρήγορα μια συνεκτική πολιτική. Και αυτό φυσικά επηρεάζει και την, ενιαία, την ιστορική αγορά και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Να πω τώρα δύο λόγια για τι συστάσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Να επαναλάβω ότι είναι υπερβολικά εστιασμένη στο βραχυπρόθεσμο πλαίσιο και αυτό θέτει ερωτηματικό σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών στοιχείων αποδοχών και των σταθερών, αν θέλετε, στοιχείων. το θέμα, θέμα του τι θα πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι που έχουν τεθεί, θα πρέπει να επιστρέφεται αυτό το άμα αυτά τα πόνους. Ένα άλλο θέμα ασφαλώς είναι τα κριτήρια της αποδόσης. Επίσης ο ρόλος της Επιτροπής Αποδοχών, ο ρόλος των ανεξάρτητων ε, ε, διαχειριστών, όλα αυτά θα πρέπει, όλα αυτά μάλλον συμπεριλαμβάνονται στις συστάσεις. Όπως ξέρετε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η ρύθμιση από 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η υποπτία θα γίνεται μέσω ετήσιων scoreboards και σχετικών αξιολογήσεων από την Επιτροπή Εργασίας των Κρατών Μελών. Όπως σας είπα, θεωρώ ότι θα πρέπει λοιπόν να πάμε λίγο παραπέρα σε σχέση με τις συστάσεις και διαπιστώνω ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ και κατά τη διάρκεια των ακρεώσεων και κατά τη διάρκεια των ε, συμβουλίων μίλησε για κατεπίγοντα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε ό,τι αφορά την πολιτική περί αποδοχών και ο Επίτροπος ε, τόνισε το ρόλο της Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής και της ε, ε, Γενικής Συνέλευσης. Αυτά λοιπόν είναι κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε και θα ήθελα να πω ότι προσπαθήσαμε μαζί με την Αρλίν Μακάφθη να διοργανώσουμε το, τις επόμενες εβδομάδες μία ακρόαση, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να τα καταφέρουμε. Ε, από ό,τι φαίνεται δεν θα τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει ο χρόνος. Η έκθεση θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στις 26 και 27 Απριλίου. Προθεσμία θα είναι η 10 Μαΐου για τις ε, τροπλογίες προκειμένου 22 Ιουνίου να λάβει χώρα η ψηφοφορία και μετά φυσικά θα περάσει στην Ολομέλεια. Αυτά λοιπόν συνάδελφοι εν είδη εισαγωγής για ένα πάρα πολύ ευρύ θέμα το οποίο χωρίς αμφιβολία θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις και ανυπομονώ να ακούσω και τα σχόλια των συναδέλφων. Ελπίζω να είναι καλή η συνεργασία μας και επικοδομητική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Βρήκε να πάρεις πρώτη το λόγο. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Τρίτη φορά συζητάμε το θέμα στην Επιτροπή τους τελευταίους μήνες γιατί προκύπτει και στην οδηγία, ε, στις τροπολογίες μάλλον για τις κεφαλαιοχικέ απαιτήσει και η Αρλίν είναι συντονίστρια. Οπότε όλοι θέλουμε να την ακούσουμε. Δεν χρειάζεται να ζητήσω συγγνώμη αν επαναλάβω κάποια σχόλια που έκανα στις δύο προηγούμενες ε, συζητήσεις. και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ευρώπη ανησυχεί το θέμα πάρα πολλούς πολίτες ε, στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε, οι φορολογούμενοι έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα για τη διάσωση των τραπεζών. Οπότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα λεφτά των μετόχων ε, για να πληρώνουν τα μπόνους ε, στα διευθυντικά στελέχη τράπεζες. Προσπαθούμε όλοι να καταλήξουμε σε μια παγκόσμια και διευρωπαϊκή συνένεση από όλες τις πλευρές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη δημιουργία πλούτου ευημερία. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πρέπει να μεριμνήσουμε ούτω ώστε να υπάρχει ευημερία. Αλλά όχι να συμπεριφερόμαστε σαν να παίζουμε στο καζίνο με λεφτά άλλων. Αυτοί που υποτίθεται ότι πρέπει να διαχειριστούν τους κινδύνους και να αρνούν τις ρηψοκίνδυνες πράξεις ε, δεν κάνουν τη δουλειά τους. Ε, και όπως είπε και ο Νιώτον ε, ε, προς τα κάτω θα πέσει το μήλο και άρα θα πρέπει βέβαια να στηρίζουμε ένα τον άλλον, να προσθέσω εδώ και σε καλές και σε κακές στιγμές, αλλά δεν έχει κατανεμηθεί ισότιμα το βάρος της κρίσης. Ε, και σε υψηλότερο επίπεδο αναφέρθηκε το θέμα των διαφόρων συμβολέων που πρέπει να επιλέξουμε βραχυπρόθεσμα, αλλά μην ξεχνάτε τι έγινε με τη Lehman Brothers οι εργαζόμενοι ήταν στενά συνδεδεμένοι με το μέλλον ε, της τράπεζας για την οποία εργάζονταν και παρόλα αυτά δεν ε, κατάλαβαν ε, τον, τον κίνδυνο. Οπότε δεν αρκούν αυτά που κάνουμε για το θέμα των αμοιβών. Οφείλουμε να εξετάσουμε την κεφαλαιοχική βάση, τη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων που θα συζητήσουμε με την Αρλίν. Επίση, πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι διαχειριστέ κινδύνου να ε, έχουν το σεβασμό που του αξίζει μέσα στου χρηματοπιστωτικού φορεί όπου εργάζονται. Επίση, μιλήσατε για την διακυβέρνηση. Ναι, ε, οι μέτοχοι και οι θεσμικοί επενδυτέ οπωσδήποτε πρέπει να διαδραματίσουν διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο ε, σε σχέση ε, με την αμοιβή για την ανάληψη κινδύνου. Με ανησύγησε αυτό που είπατε για την ισορροπία ανάμεσα στα μπόνους και τη βασική αμοιβή, το βασικό μισθό. Ε, την περασμένη εβδομάδα διάβαζα ότι ε, σαφώς κάποιοι κάνουν φοβερές προσπάθειες εγκαταλείπτοντας ε, το, τα μπόνους τους και ότι αυτό ε, θα βοηθήσει τους φορολογούμενους. Άλλοι πάλι αποφάσισαν να μειώσουν τους μπόνους αλλά να αυξήσουν σημαντικά το βασικό μισθό. δεν πιστεύω ότι αυτό είναι πιο βιώσιμος τρόπος διεύθυνση μιας επιχείρησης. Χρειάζεται κάποια αμοιβή όταν αναλαμβάνει κάποιος κίνδυνο αλλά χρειάζεται και μέτρο. Ε, οπότε δεν είμαι σίγουρο ότι είναι καλύτερο να αυξήσουμε το μισθό για να μειώσουμε τον πόνους. Ε, κάτι άλλο τώρα. Είναι παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά αυτή στην οποία δραστηριοποιούμαστε και δεν μιλάμε μόνο για χρηματοπιστωτικούς φορείς εγχώριους ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουμε, φτιάχνουμε μέτρα και κανόνες χωρίς όμως να κοιτάζουμε λίγο παρά έξω τι συμβαίνει στον κόσμο. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι κάνει το FSB και κάποια κρατημέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες. Όπως σας είπα στη συζήτηση για τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει ε, που ε, βρίσκεται στη βάση του συστήματος ε, αμοιβών, ας δούμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τι θέλει να κάνει ο κύριος Σαρκοζή στη Γαλλία. Ίσως κάποιοι να πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ, Κάρλ Χάγκλουντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση σε αυτό το θέμα ε, και πριν από 10 χρόνια είχαμε πει ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι για να ρυθμίσουμε το σύστημα. Είναι κρίμα που δεν ε, κινηθήκαμε ταχύτερα για να προλάβουμε αυτή την κρίση. Ε, ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξουν κάποιοι σοφότεροι σε κάποιους κλάδους, σε κάποιες οικονομίες σχετικά με την ανάληψη κινδύνου. Έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να δεχθούμε ότι επί της αρχής πρέπει να γίνουν συστάσεις και να αναλυθούν δράσεις. Και το βλέπουμε αυτό τις εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ταυτόχρονα ε, πρέπει να χαρακτηρίζονται οι δράσεις μας από ισορροπία. Ε, η οδηγία για τα εναλλακτικά ταμεία επενδύσεων. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό με αυτά που συμβαίνουν εδώ, διότι υπάρχει μια ένα λαϊκιστικό, αν θέλετε, θεματολόγιο που μας ε, ανησυχεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση προς τους πολιτικούς ε, για να κινηθούν με πυγμή ε, σε τέτοια θέματα και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ε, και ξέρετε όμως ε, θα πρέπει να κάνουμε και τη διαφοροποίηση με το θέμα των ελεκτικών επενδυτικών ταμείων ε, γιατί πρόκειται για διαφορετικές δραστηριότητες και θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά τι συστάσεις θα κάνουμε. Επίσης είναι γεγονός ότι η επιχειρηματική κουλτούρα στην Ευρώπη είναι διαφορετική σε σχέση με αυτή που επικρατεί στη ΣΥΠΑ οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη. Καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Επίσης, είναι καλό να έχουμε κατά νου ότι ενέχεται ένας κίνδυνος, ε, συστημικός κίνδυνος ε, για τον κλάδο, οπότε δεν πρέπει απερίσκεπτα να αναλαμβάνονται κίνδυνοι. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμιστεί και το θέμα των αμοιβών επίσης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ξέρουμε γιατί υπάρχει ένα σύστημα αμοιβών. Πριν ε, το καταργήσουμε, το σύστημα αμοιβών δεν δημιουργήθηκε μόνο για να έχουν πολλά λεφτά οι διοικητές των τραπεζών. Ε, είναι αποσκοπή ε, στην δημιουργία ευημερίας στην κοινωνία μας γενικότερα. Οπότε πρέπει να έχουμε μια ισορροπία Και όπως ε, είπε τώρα η συνάδελφο, ε, δεν είναι πολύ καλύτερο να αυξήσουμε το μισθό για να μειώσουμε ή να καταργήσουμε τα μπόνους. Δεν είναι απαραίτητα καλύτερο. Θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη πριν να αποφασίσει η Επιτροπή να ρυθμίσει ε, τον τομέα αυτό. Και το βασικό είναι να ορίσουμε ποιο είναι υπεύθυνο γιατί και επίσης ότι θα υπάρχουν επαρκείς πόροι για το σύστημα ε, που θα θεσπίσουμε και ορισμένες φορές είναι κακό το να ρυθμίζουμε τόσο λεπτομερώς αυτά τα ζήτημα. Πάντω είναι επικοδομητική και λογική η προσέγγιση του εισηγητή αλλά ε, μην ξεχνάμε πόσο πολυδιάστατο είναι το ζήτημα. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο ή τον εισηγητή για την πάρα πολύ σωστή προσέγγιση που υιοθέτησε για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε το εξή. Το θέμα αυτό θα το συζητούσαμε αν δεν είχε προκύψει η οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι οι οικονομικοί κανονισμοί σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, τη διαφάνεια, θα ήταν επαρκής σε περίπτωση που δεν είχε προκύψει η κρίση. Αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εξέβρεση μηχανισμών για να αντιμετωπίσουμε τα αυτά εν και της κρίσης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να διαχωρίσω την ε, διαχείριση βάσει της ε, κατάστασης της αγοράς από την οικολογική κατάσταση που προέκυψε. Θα πρέπει να καλύψουμε όλο το φάσμα των πτυχών αυτών Η ρύθμιση λοιπόν θα πρέπει να περιοριστεί θα πρέπει να περιορίσει τη βράχη πρόθεσμη επικίνδυνη συμπεριφορά ε, στις αγορές ε, και τις σχετικές ε, αποδοχές. Αυτό αποτελεί μια παθολογική κατάσταση η οποία θα πρέπει να αποφευθεί. Κάτι άλλο το οποίο αποφασίζεται στην πραγματικότητα. Αν κάποιος χρησιμοποιεί κρατικές επιδοτήσεις, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι δημόσιες αρχές βασίζουν την πολιτική αποδοχών σε πολύ διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός είναι παθολογικής φύσεως αν διατηρηθεί έτσι χρησιμοποιώντας ε, τις κρατικές ενισχύσεις, τις κρατικές επιδοτήσεις, θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική ρύθμιση. Θα ήθελα όμως να σας καλέσω να διαχωρίσουμε τις επιχειρήσεις αυτές που βρίσκονται στο όριο, αν θέλετε, από την φυσιολογική αγορά, όπου δεν έχουν προκύψει κίνδυνη, δεν έχει προκύψει κρίση. Δεν θα πρέπει να τους επιβληθούν, δηλαδή επιπρόσθετες, ε, επιπρόσθετοι περιορισμοί. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία τώρα. Η εποπτεία γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη όταν αντιμετωπίζουμε μία απειλή. Συμφωνώ με όσους ανέφεραν ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε με μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί σχετίζεται και με θέματα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μακάρτη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πολλά ήδη υπόθηκαν και ε, πολλά σωστά υπόθηκαν σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, το οποίο ασφαλώς δεν αφορά μόνο τον τραπεζικό κλάδο. Χαίρομαι που ο εισηγητής μας και ο συνάδελφος ε, όρισε ένα συνεκτικό τομέα για να εξετάσουμε τις προτάσεις αυτές. Ξέρω ότι δεν είχαμε χρόνο για ακρόαση, αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε λάβει τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, γιατί είναι περίπλοκος ο κλάδος αυτός. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε προτάσεις ε, και να υποβάλουμε προτάσεις περιοριστικές. Θα πρέπει να θέσουμε κάποιες γενικές αρχές, τις οποίες όλες οι πολιτικές και όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρούν. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποιος είναι ο βασικός μας στόχος. Όχι, βασικ... όχι βέβαια τα ηθικά θέματα τα οποία συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι θα πρέπει να τα θίξουμε. Γιατί αυτό ήταν πολύ σημαντικό στην τρέχουσα κρίση. Δεν τηρήθηκαν κάποιοι ιδεολογικοί κανόνες από τις αγορές, αλλά ο βασικός στόχος είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει η προστασία και η βελτίωση της σταθερότητας του οικονομικού μας συστήματος. Αυτός θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος. Και γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι οι αρχές αυτές, η καθιέρωση αρχών είναι σωστός τρόπος. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα πρέπει να γίνει. Γιατί κάποιοι μέτοχοι στην κρίση, αμα, είδαμε ότι στην κρίση την παρούσα είδαμε ότι οι μέτοχοι σε πολλές περιπτώσεις κοιμόντουσαν. Ή όχι μόνο κοιμόντουσαν, αλλά είχαν συμφέρον να αναλευθούν μεγαλύτερη κίνδυνη. Γιατί αυτό θα σήμαινε μεγαλύτερα κέρδη για αυτούς. Και θεωρώ ότι και οι επενδυτές θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των αποδοχών. Όχι ότι θα πρέπει να προδιαγράφεται φυσικά το επίπεδο των αποδοχών. Υπάρχουν, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, πόσο ξέρω, φόρουμ ε, μετόχων και των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό ως μία λύση. Και σε ό,τι αφορά φυσικά και οι επιτροπές αποδοχών. Χρειάζεται πολύ περισσότερη διαφάνεια, γιατί όσο πιο πολύ διαφάνεια υπάρχει, τόσο πιο πολύ διαφωτίζονται οι πολιτικές των εταιριών σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις πρακτικές υψηλού κινδύνου και την κοινωνική τους ευθύνη. Ακούσαμε επίσης η κερδοφορία ασφαλώς δεν είναι ε, σε καμία περίπτωση κάτι το εσφαλμένο. Αυτό οθεί και την οικονομία άλλωστε. Αλλά θα πρέπει να ορίσουμε ότι η πολιτική αποδοχών δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να επιβραβεύει την αποτυχία. Και αναφέρθηκε ότι φέτος ε, τα στελέχη δεν θα πάρουν τα μπόνους τους. Αυτό το αναφέρουν λες και μας κάνουν χάρη. Γιατί να πάρουν όμως μπόνους στη στιγμή που ε, υπήρξαν τέτοια τεράστια προβλήματα. Θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει λοιπόν η κουλτούρα και θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε ό,τι αφορά την πολιτική των αποδοχών στις χρηματοπιστωτικέ ε, υπηρεσίε. Και γι' αυτό χρειάζονται σωστέ προτάσει. Και πάλι τονίζω ότι προτιμώ μια προσέγγιση επί της αρχής, γιατί αν επισέλθουμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να ανταποκριθεί στις ανάγκες και των 27 κρατών μελών. Δεν θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε το κέρδος, θέλουμε, δεν θέλουμε όμως την δικοποίηση του κέρδους και ε, κοινωνικοποίηση, αν θέλετε, δημοσιοποίηση των απολειών, των ζημιών. Και συμφωνώ ιδιαίτερα με όλα όσα μας θα ανέφερε ο εισηγητής. Ο Σβέν. Ευχαριστώ. Σύντομα, να πω ότι μου κάνουν εντύπωση κάποιες από τις παρατηρήσεις που, από τις που έγιναν. Είπατε ότι η συζήτηση αυτή διέπεται από τον λαϊκισμό και ότι διακυβεύω την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα πρέπει να σας πω ότι η ανάλυση της κρίσης καταδεικνύει με σαφήνεια ότι υπήρξαν υπερβολικά κίνητρα για υπερβολική ανάληψη κινδύνου. Και θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για να αποφευθεί αυτή η διαμόρφωση εκ νέου των κινήτρων αυτών σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να αναλυφθεί δράση. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Δεν διακυβεύουμε έτσι την ε, ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της, ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Γιατί μάθαμε από την κρίση ότι οι αποφάσεις για τις αποδοχές που ελήφθησαν από τις επιτροπές και από το Εποπτικό Συμβούλιο δεν ήταν προς το συμφέρον των μετόχων ούτε προς το συμφέρον της γενικότερης οικονομίας. Εξετάζοντας λοιπόν τις αρχές οι οποίες ε, α, αναφέρονται στο έγγραφο της Επιτροπής, είναι μάλλον ασαφείς και τέτοιες ασαφείς ε, συστάσεις δεν αξίζουν καν το χαρτί που έχουν γραφτεί. Θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς. Αν ε, αναφέρουμε ότι χρειαζόμαστε πολιτικές οι οποίες θα εστιάζονται το μακροπρόθεσμο α, επίπεδο θα πρέπει να δούμε το μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό κύκλο. Στη Γερμανία υπάρχει μία νέα νομοθεσία η οποία προβλέπει πλέον τρία χρόνια. Τρία χρόνια όμως δεν επαρκούν για να αποδείξουν ότι, για παράδειγμα, έχει αναλυφθεί υπερβολικά μεγάλος κίνδυνος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό το ευέλικτο στοιχείο, το μεταβλητό στοιχείο των αποδοχών, απλά με τους σωστούς όρους. Η δεύτερη αρχή είναι σαφής. Αν υπάρχει ένα τέτοιο μεταβλητό στοιχείο, θα πρέπει να είναι και αρνητικό και θετικό, όχι μόνο θετικό, και κατά τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει σαφής περιορισμός του μεταβλητού στοιχείου των αποδοχών. Για παράδειγμα, σε ύψος 25% του συνόλου της αμοιβή. Θα ήθελα να τονίσω όμως ότι το βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να εξαγάγουμε ως μάθημα από την κρίση δεν είναι τόσο πολύ το επίπεδο των ε, αποδοχών αλλά το να σταματήσει αυτή η κουλτούρα της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων σε ό,τι αφορά την πολιτική των αποδοχών. Οι κανόνες λοιπόν που θα πρέπει να τεθούν στα πλαίσια της ε, έκθεσης Μακάρθη και Ελκαντράουι θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί και συγκεκριμένοι, όχι ασαφείς. Θα πρέπει να διδαχθούν από τα συμπεράσματα της κρίσης, από τα παθήματα της κρίσης η Πρόεδρος. Επειδή ο εισηγητής ε, πρέπει να μεταβεί στην Επιτροπή Μεταφορών να παρουσιάσει άλλη ε, έκθεση, αλλά θα συζητηθούν, ε, θα, μάλλον θα σημειωθούν οι υπόλοιπε εισηγήσει. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον Ζαν Κοιτάξτε, Πρόεδρε, για αυτό το θέμα των αμοιβών ε, ε, υπάρχουν πολλά ανάμεικτα συναισθήματα και θα το ξαναζητήσουμε το θέμα. Μιλάμε για εικονική και πραγματική οικονομία. Το πρώτο πρέπει να μας απασχολήσει είναι αν νομιμοποιούνται τόσο υψηλέ αμοιβέ σε σχέση με τη συνεισφορά αυτών των ατόμων στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτό το θέμα ε, των χρηματοπιστωτικών φορέων έχει ως αποτέλεσμα οι καλύτεροι μηχανικοί, οι καλύτεροι μαθηματικοί, οι καλύτεροι επιστήμονες ε, προτιμούν να κάνουν τους traders και να μαζεύουν λεφτά παρά να φτιάχνουν δρόμους, γέφυρες ή ανανεώσιμες ενεργειακές ε, πηγές. Μα αυτό είναι το πραγματικό θέμα, όχι μόνο να λέμε πόσα βγάζουν. Τέλος πάντων, ε, στη, στην τράπεζα, γιατί ξέρω τι λέω, στη Société Générale, ε, γαλλική τράπεζα ε, ο πρώην ε, ε, πρόεδρος ήταν ο 30ος μισθός. Δηλαδή δεν είχε αυτό τον υψηλότερο μισθό. Οι φυστάμενοι του είχαν τον υψηλότερο μισθό που ανελάμβαναν κινδύνους για μέσω μακροπρόθεσμα και όταν φτάνουν παίρνουν αυτό το παχυλό μπόνους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω εγώ να καταστραφούν όλοι αυτοί που είχαν τα υψηλά μπόνους, Μία, αλλά να υπάρχει κάποιο μέτρο ε, ανάμεσα στην αμοιβή και την συμβολή στην οικονομία αυτού του ατόμου. Λέμε ότι α, θα καταρακωθεί η οικονομία. Ε, μα τι, ε, ε, δείτε στο Ντουμπάι τι έγινε ας πούμε με τη φούσκα. το ίδιο θα γίνει και με τα hedge funds, τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου. Κάνιν. Η κυρία Βόρτμαν Κόλλε. Ναι, λυπάμαι, Πρόεδρε, που δεν ήμουν παρούσα στην παρουσίαση του εισηγητή. Θα ήθελα όμως να απαντήσω σε κάποιες από τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως εκπρόσωποι του λαού, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό των μπόνους, ε, γιατί οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες υπερβολικές ε, αμοιβέ, τέτοια υπερβολικά μπόνους σε τράπεζες που πτωχεύουν και όπου σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να επανέρχεται το φαινόμενο αυτό. Να υπάρχει απειλή τέλο πάντων ε, ε, επανόδου και επανεμφάνισης τέτοιων ε, φαινομένων. Και όλα αυτά φυσικά συνέβαλαν και στην κρίση, το ξέρουμε. Και αναγκαστήκαμε με δημόσιο χρήμα να σώσουμε τις τράπεζες μας. αλλά πρόεδρε δεν πιστεύω ότι θα διορθωθεί η κατάσταση από μόνη Θα πρέπει, όπως και σε άλλες περιπτώσει να υποβάλουμε προτάσεις για ρυθμίσεις. Θεωρώ ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν πολλές καλές ιδέες σε ό,τι αφορά τις αρχές οι οποίες ισχύουν και στην Ολλανδία, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ισότιμο επίπεδο, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τα μπόνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη για το επίπεδο των αποδοχών αυτών, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τις αρχές που θα πρέπει να τηρούνται από τους Ευρωπαίους εποπτικούς οργανισμούς, όχι μόνο από τις, εθνικούς, από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Και εδώ συμφωνώ με τους συναδέλφους να προσέξουμε να μην ε, καταλήξουμε τελικά σε μια υπερβολικά λεπτομερή νομοθεσία, σε μια υπερβολικά ε, λεπτομερή ρύθμιση, γιατί δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η φορολογία σε ό,τι αφορά τις αποδοχές αυτές που έχει εισηχθεί ή πρόκειται να εισηχθεί σε κάποιες ε, χώρες. Δεν αποτελεί και αυτή η λύση, γιατί δεν θα περιορίσει την συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, ανάληψης υψηλού κινδύνου και σε αυτόν τον κλάδο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα level playing field, ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ, ο Έντουαρτ. Πριν μιλήσουμε για τις αστρονομικές αμοιβέ των μεγάλων στάρ, των τραγουδιστών, των ποδοσφαιριστών. Φαίνεται ότι είμαστε θεότρελοι, αλλά το ίδιο γίνεται και με την χρηματοοικονομική αγορά. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το λόγο, όπως είπε και ο κύριος Γκοζές, λυπάμαι διότι τα καλύτερα ε, μυαλά αντί να ασχοληθούν με τη μηχανική ή αλλού ασχολούνται με τον χρηματιστηριακό τομέα εξαιτίας των αμοιβών και αυτό φαίνεται και από τα πανεπιστήμια μας. Ε, ορισμένες σχολές ε, δύσκολα ψαρεύουν φοιτητές ενώ οι οικονομικές σπουδές πάνε πολύ καλά. Το ζήτημα είναι γιατί καταβάλλονται αυτοί οι μισθοί και όταν σκάσει η φούσκα βλέπουμε ότι υπάρχει αγώνας ε, αγώνας τρεξίματος προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ διαφορετικά όταν, όταν σκάσει εντελώς η φούσκα ασχολούνται οι άνθρωποι με άλλα, όπως κυπουρικοί. Η ουσία είναι ότι καταφέραμε να βρούμε διέξοδο σε μια βιομηχανία η οποία δεν τα κατάφερε καθόλου καλά εξεράγει και μετά ο φορολογούμενος ήταν αυτός ο οποίος έπρεπε να καταβάλει το τίμημα. Αυτή ήταν η ουσία. Αν το δούμε υπό αυτή την οπτική γωνία, θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο αυτή η πρακτική οδηγεί σε αυτό το ξέσπασμα, σε αυτή την εφορία και τον, ε, την υπερβολική ανάληψη κινδύνων. Αυτό είναι ένας ουσιώδης λόγος. Ο άλλος λόγος ίσως είναι ο λαϊκισμός, ίσως είναι λαϊκισμός. Αλλά τι αισθάνονται οι άνθρωποι, διότι είναι οι φορολογούμενοι και ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναζητήσει τα χρήματα, να τα βγάλει από την τσέπη του για να επιδοτήσει και να βρει διέξοδο στον χρηματιστηριακό τομέα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο φορολογούμενος καταβάλει το τίμημα όμως αυτού του σχεδίου διάσωσης και γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε κανόνες που να είναι αποδεκτοί στο γενικό κοινό και σε όλους εμάς. Όλα. Όλα. Sorry, I was a bit late. Λυπάμαι που άργησα, αλλά από τις 8 το πρωί βρίσκουμε στο αεροδρόμιο. Νομίζω ότι βεβαίως πρέπει να αντιδράσουμε. αλλά θα ήθελα να πω ότι ίσως θα πρέπει να είμαστε πιο εξισορροπημένοι και θα ήθελα να το πω προς το συναδελφό μου, τουλάχιστον στη χώρα μου γίνονται συζητήσεις και ο προτινόμενος κανονισμός δεν στοχοθετεί μόνο τις τράπεζες που δεν τα κατάφεραν καθόλου καλά και δεν συμπεριφέρθηκαν καλά, αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία αύξηση των συνολικών μισθών, διότι το σύστημα αμοιβών, το σύστημα μπόνους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν ισχύει ένας κανόνας για τα πάντα που να καλύπτει όλες τις καταστάσεις. Ελπίζω λοιπόν να φτάσουμε σε μια εξισορροπημένη προσέγγιση. Δεν πρέπει να είμαστε λαϊκιστές, αλλά υπάρχει μεγάλη, μεγάλη δυσαρέσκεια από το κοινό. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Πρόεδρος, και εγώ χωρισμένα σχόλια. Μιλήσαμε για τους κινδύνους και μπορούμε να ζητήσουμε από τους επόπτες να ορίσουν κανόνες σε σχέση με τη ρευστότητα, το κεφάλαιο και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι προστατευόμαστε και εμείς και τα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα από τους κινδύνους. Αλλά μιλάμε για δεοντολογία ή πολιτισμικό υπόβαθρο. Εν πάση ε, για ό,τι και να πρόκειται, δεν ε, εναποτίθεται πια στους επόπτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσουμε κανόνες συμπεριφοράς. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτές οι υποδείξεις που αφορούν διάφορα φόρα, διαρθρωτικά μέτρα ή διοικητικά συμβούλια, όλα αυτά μπορούν να ασκήσουν πίεση σε πολιτισμικό επίπεδο. Είναι καλές κινήσεις, αλλά νομίζω ότι φτάσαμε στο στάδιο όπου ίσως αυτό να μην αρκέσει πλέον για ορισμένα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως οι τράπεζες και υπάρχει μεγάλη διαφορά αν ε, κανείς είναι σε μία ε, επιχείρηση που έχει μπει στο χρηματιστήριο σε σχέση με μία επιχείρηση η οποία και να μην πάει καλά δεν πρέπει να διασωθεί γιατί πολλές φορές ο φορολογούμενος είναι αυτός που καταβάλει το αντίτιμο και ίσως θα πρέπει να αντιταχθούμε στο κέρδος του χρηματοπιστωτικού τομέα για να δούμε πού έγκυται το λάθος. Αν γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, 20 χρόνια πριν, το χάσμα μεταξύ των πλέον πλουσίων και των λιγότερο πλουσίων ήταν πολύ μικρότερο από το σημερινό και υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του, της αναπτυξιακής πορείας αυτού του χάσματος και της, ε, του, της αναπτυξιακής πορείας του πιστοτικού συστήματος. Άρα υπάρχουν ε, πιστώσεις πολύ ψηλότερες σε ατομικό επίπεδο. Γι' αυτό το χάσμα γίνεται όλο ένα και πιο μεγαλύτερο σε σχέση με αυτούς που επινόησαν αυτό το σύστημα και απότοκο ε, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να χορηγήσουμε μεγάλο τμήμα αυτών των πιστώσεων συμμετρικά. Ίσως θα έπρεπε να απαλλαγούμε από αυτή την κατάσταση του να έχουμε αυτό το υψηλό, το μεγάλο χάσμα μεταξύ πλουσίων και υπολείπων, ιδιαίτερα σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα έγινε λόγος για ισολογισμούς και όλα τα σύναφη, αλλά και ως φιλελεύθερη μένω άναυδη και θεωρώ ότι μερικά ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν. Φτάνει πια. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο και φτάσαμε και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή ως προς τα κινητά τηλέφωνα και τις χρεώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι και ως φιλελεύθεροι θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στους επόπτες και να τους πούμε χειριστείτε το. Δεν πρόκειται μόνο για τα μπόνους, αλλά για το συνολικό σύστημα αμοιβών. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι προτάσεις που θα ανακύψουν και στο CRD και σε αυτό το πλαίσιο μεταξύ αυτών που θα πρέπει να ε, οριστούν εναπόκειται και αυτό το θέμα, δηλαδή η πολιτική αμοιβών του χρηματοπιστωτικού τομέα και ιδιαίτερα των υψηλόβαθμων στελεχών. Δεν ισχύει ένα μέτρο για τα πάντα. Θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση, όχι μεταξύ των εισηγμένων και του χρηματοπιστωτικού τομέα υπηρεσιών, αλλά και μέσα στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού καθεαυτού. Αυτά είχα να πω και θα επανέλθω στον Ούντο, ο οποίος έχει το λόγο εξ του εισηγητή, για να συνοψίσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αντικαθιστώ τον εισηγητή της ομάδας μας, τον κύριο Ελκαντράουι. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή αλλά να ευχαριστήσω και την κυρία Πρόεδρο για τις δηλώσεις που έκανε σε ό,τι αφορά τους σαφείς κανόνες που θα πρέπει να υπάρχουν ε, στην αγορά. Νομίζω ότι οι δύο εισηγητές που είναι υπεύθυνοι για τα θέματα αυτά, ο κύριος Ελκαντράουι, αλλά και η κυρία Μακάρθη, έκαναν σαφές πόσο ε, έντονα θα παρακολουθήσουν το θέμα αυτό. Και όντως, εμείς ε, ως Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων θα πρέπει να εξαγάγουμε ένα μάθημα από την οικονομική κρίση. Γιατί η οικονομική κρίση την πληρώνει κάθε μέρα ο κόσμος. Ο κόσμος που χάνει το, τη θέση εργασία του, που δεν βρίσκει καινούργια δουλειά και διεθνώ πάσχουμε. Και θα πρέπει φυσικά να καλέσουμε τα κράτη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το συζητήσαμε σήμερα, αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριφερθούν με υπεύθυνο τρόπο προκειμένου να καταλήξουμε σε μια υγιή ισορροπία. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, απλά να πω ότι ο συνάδελφος ανυπομονεί να ακούσει τις απόψεις των συναδέλφων και ελπίζει να υπάρξει καλή συνεργασία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Όπως είπε και ο εισηγητής, η εξέταση της ε, Επιτροπής προγραμματίζεται για τις 26 Απριλίου, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 10 Μαΐου, 1 Ιουνίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 22 Ιουνίου, προκειμένου να περάσει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Ευχαριστώ λοιπόν ε, τους συναδέλφους πέρα στη συνεδρίασης και θα ξεκινήσουμε στις 9 αύριο το